γιατί εκεί σε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

Good morning, ladies and gentlemen. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ε, λυπούμε που σας έκανα να περιμένετε, αλλά είχα κάπου μια άλλη συνεδρίαση. Αυτή η συνεδρίαση βέβαια είναι ιδιαίτερη σημασία για μένα. Έχω προετοιμάσει μια ομιλία για σήμερα το πρωί. Πολύ μακρά. Και είσαστε ευτυχείς φαντάζομαι, ε, θα με ακούσετε. Λοιπόν. Διαβολίζουμε μακρά, αλλά προτιμώ να σας πω μόνο δύο λόγια ενώπιον ημών. Πιστεύουμε στην Ευρωπαϊκή μας Ένωση. Εγώ πιστεύω απόλυτα σε αυτή. Πριν από μια εβδομάδα ήμουνα στην Πράγα και μίλησα για την Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί, που ενδιαφέρονται και εκεί πάρα πολύ, θα πρέπει να σας το πω. Στο Κοινοβούλιο πρέπει να κάνουμε κάτι βέβαια για την Προεδρία της χώρας αυτής, αλλά η χώρα, οι πολίτες ενδιαφέρονται πάρα πολύ. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Υπάρχουν κάποια προβλήματα ίσως. Από την άλλη μεριά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εσάς σας χρειαζόμαστε για να ενημερώνετε τους πολίτες για όλα όσα λαμβάνουν χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδίως γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όσον αφορά τη συμμετοχή όλοι μας χάσαμε τις εκλογές. 40% συμμετοχή δεν είναι επαρκή. Είναι βέβαια πάντα καλύτερη από ό,τι για το Αμερικανικό Κογκρέσο που έχουν 37% αλλά για μας δεν αρκεί αυτό γιατί η δημοκρατία είναι το έργο μας. Πρέπει να είμαστε πιο δημοκρατικοί. Δεν υπάρχει δυνατότητα βέβαια να επικοινωνήσουμε με τους πολίτες χωρίς εσάς τους ε, δημοσιογράφους. Στο διαδίκτυο, στον γραπτό τύπο, στο ραδιόφωνο στην ε, τηλεόραση. Τέσσερις κατηγορίες λοιπόν, στις οποίες σας εργαζόμαστε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αλλιώς χάνουμε την επαφή με τους πολίτες. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή εδώ η συνεδρίαση είναι ένα μήνυμα για τη συνεργασία μας, για την αναγκαιότητα να είμαστε σε επαφή ημέν με τους δε. Μπορώ να σας πω ότι μετά την επίσκεψη στην Πράγα, ότι είναι σίγουροι ότι θα λειτουργήσει η συνθήκη της Λισαβόνας το επόμενο έτος, γιατί δεν είναι εύκολο αυτό. Δεν είναι εύκολο για όλες αυτές τις χώρες μέλη που θέλουν ε, Ακούνε βέβαια τι προτάσει τη Τσεχική Δημοκρατία. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αλλά πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Ξέρετε πόσο σημαντικό αυτό. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί. Έναντι των πολιτών. Να ανταποκριθούμε στο πρόβλημα τη ενεργείας. Να ανταποκριθούμε στα προβλήματα τη ε, <clears throat> με φυσικό αέριο με ηλεκτρική ενέργεια, με τα προβλήματα της μετανάστευσης, κλιματολογικές αλλαγές, δημογραφικά προβλήματα και ούτω καθεξής. Είναι μια πολύ καλή ημέρα σήμερα γιατί έχουμε το δεύτερο βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους δημοσιογράφους. Έχουμε τέσσερις κατηγορίες όπως σας είπα, αλλά καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αντιπρόεδρο κυρία Ρώδη Κράτσα Σαγκαροπούλου για την έντονη υποστήριξή της. Πού είσαι? Probably she will come. Δεν είσαι ακόμα εδώ. Θα έρθει. Βέβαια. Ε, μια άλλη συνάδελφος. Η κυρία Κοχμερίν, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Κοιτάω το όνομά σας για να μην το προφέρω λάθος. Συνάδελφος Μόρτον Λόκενκάρτ, που ήταν ε, στην Προεδρία της συνάντησης της ε, Τελεσκέψης το πρόεδρο της ε, Διεθνούς Ένωσης Δημοσιογραφίας, να ευχαριστώ Φραντσέσκα Ράτη, από τη Γενική Γραμματεία, ε, ε, Διεύθυνση συγγνώμη, που οργάνωσε αυτή την ε, απονομή του βραβείου. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που συμμετέχατε στην, ε, στο διαγωνισμό αυτό. Πρώτη φορά δώσαμε το βραβείο αυτό πέρσι, τώρα είναι η δεύτερη φορά. Τώρα ας αρχίσουμε λοιπόν τώρα την επίσημη τελετή, γιατί όλοι έχουμε πολλές δουλειές, και εσείς και εγώ. Και εσείς έχετε πολλά τόσα νέα πρέπει να συλλάξετε και να μεταδώσετε. Ας αρχίσουμε λοιπόν, κυρία μου, αμέσως. Αρχινήχω το πρώτο φάκελο εδώ. Είσαστε έτοιμοι. Fantastic. Θαυμάσια. Όλοι είναι έτοιμοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, τα γελιά μου τα ξέχασα, αλλά εντάξει, θα διαβάσω χωρίς γελιά. Διαβάζω και χωρίς γελιά, φαντάζεστε. Ε, στην κατηγορία του γραπτού τύπου το βραβείο χωρίς στην Ίνες Πόσε από τη Γερμανία για το άρθρο πώς αναδυνώνεται η Ευρώπη. Παρακαλώ. Congratulations. It's for you. The... Συγχαρητήρια. Το άρθρο από την Ίνες Πόσε λέει... With brilliant photographs η Κρητική Επιτροπή είναι πάρα πολύ ενημερωτικό. Ορίστε, για σας. Μαζί και τώρα μόνοι σας. Αυτά. Συγχαρητήρια. Well, fine. Maybe I should, I should smile much more. Well, Ίσως να χαμογελάω για τις φωτογραφίες. Σας παρακαλώ, μπορείτε να μας απευθύνετε δύο λόγια. Επιτρέψτε να μιλήσω στα γερμανικά. Ναι, καταλαβαίνω, λέει ο πρόεδρο, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι μέλη τη Κριτική Επιτροπή, Θα ήθελα καταρχά να σα ευχαριστήσω όλου ε, για την τιμή που μου κάνετε και να, και να συγχαρώ όλου του ε, νικητέ όσου απονεμηθεί το βραβείο. Είναι πολύ μεγάλη τιμή που βρισκόμαι στην καρδιά σχεδόν της Ευρώπης. Έχω στην ε, ζωή μου ασχοληθεί ιδιαίτερα με τις ε, διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης, την Νότια Πολωνία, την Ιρλανδία, την, ε, τα σύνορα μεταξύ Ρουμανίας και, Βουλγαρίας. Έχω κινηθεί και πρέπει να πω ότι μπόρεσα να παρακολουθήσω τις μεγάλες αλλαγές που διαγράφονταν στη μεγάλη ευρωπαϊκή σκηνή. Θα ήθελα λοιπόν πολύ σύντομα να μιλήσω για πρωτοπόρους και για περιφέρειες. Η επανένωση της Γερμανίας και η διεύρυνση προς Ανατολάς της Ευρώπης ε, ε, ε, προκάλεσαν μεγάλες κινήσεις πληθυσμών από τα, μεταξύ των παλαιών και νέων κρατών πολιτών οι οποίοι έρχονταν και για νέες εμπειρίες αλλά πάνω απ' όλα για νέες ευκαιρίες στη ζωή τους και το φαινόμενο αυτό εγώ το βίωσα στην ε, γέφυρα πάνω στο Ιδούνευη που χωρίζει την, που ενώνει μάλλον τη Βουλγαρία με την ε, Ρουμανία. Ήμασταν ε, μακριά από το Βουκαρέστι, περίπου 70 χιλιόμετρα. Σε ένα σημείο λοιπόν της Μεθορίου, όπου είδαμε ότι περνούν ε, καθημερινά οι εργαζόμενοι, οι, οι φοιτητές ακόμη, όπως μια Πολωνίδα η οποία πηγαίνει από τη μία μέρα, κάθε μέρα να εργαστεί από τη μία πλευρά στην άλλη. Όταν είδαμε ότι η μία χώρα η οποία ήταν φτωχή παλαιότερα, όπως η Ιρλανδία, έστελνε εργαζόμενους ή λάμβανε μάλλον εργαζόμενους πλέον από ένα νεότερο φτωχό κράτος ε, και όταν είδαμε ότι η λαμβανε μαλλον εργαζομενου πλεον απο ενα νεοτερο φτωχο κρατο και οταν ειδαμε οτι η έννοια της γειτνίασης ήταν μόνο λόγια στα στόματα των ε, πολιτικών, ενώ αποτελούσε βίωμα για τους κοινού πολίτες. Εκεί όπου ο μετανάστης, είτε προσπαθούσε την οικονομική του και ε, την, την καθημερινή του ζωή να βελτιώσει. Και εκεί είδαμε ότι οι περιφέρειες πολλές φορές έχουν να αντιμετωπίσουν πολύ δύσκολες συνθήκες σε διάφορες απομακρυσμένες περιοχές όπως την Βόρεια Ισπανία, την Νότια Ιταλία, την Ανατολική Γερμανία που χάνουν καθημερινά πολίτες και κυρίως νέους πολίτες. Και εκεί υπάρχει και χαμηλό επίπεδο γεννητικότητας. Έτσι λοιπόν ε, βλέπουμε ότι μακροπρόθεσμα γυράσκει ο πληθυσμός στις περιοχές αυτές ε, και ότι θα πληγούν μακροπρόθεσμα και άλλες περιφέρειες της Ευρώπης, όχι μόνο αυτές οι πιο φτωχές, που θα παρουσιάσουν ε, πολύ σύντομα και σε ρήγνωση του πληθυσμού, εάν δεν έρθουν νέοι μετανάστες έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και γύρανση. Θα είμαστε σε λίγα χρόνια, κατά δέκα χρόνια, πιο ηλικιωμένοι από την τωρινή γενιά της Ευρώπης, κατά μέσο όρο δηλαδή. Έτσι, υπάρχει ο κίνδυνος η Ευρώπη να ε, χάσει το κεντρικό της ρόλο στην διεθνή σκηνή και να μετατραπεί σε, πολι... σε περιφερειακή μονοδύναμη. Εγώ ελπίζω ότι αυτό δεν θα υλοποιηθεί. Ελπίζω ότι αυτή μεταναστευτική... αυτές οι μεταναστευτικές ροές θα αποτελέσουν και ε, πόλο ενδυνάμωσης της Ευρώπης και χάρη στην συμπεριφορά που θα τηρήσουμε απέναντι στο στο κλίμα και τις κλιματικές αλλαγές και στο περιβάλλον μπορούμε να αποτελέσουμε έναν ε, πόλο σταθερότητας και όχι ε, αποτυχίας. Μπορεί η Ευρώπη με τις πολλαπλές πολιτιστικές παραδόσεις που έχει να προβάλλει να δείξει πώς μπορεί κανείς ε, να συμβιώσει αρμονικά μαζί με τους άλλους. Μπορεί κάποιοι να είναι καλύτερα εξοπλισμένοι από κάποιοι άλλοι, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε μαζί όλοι πρωτοπόροι και στην ε, εξέλιξη τη δημογραφική, αλλά πάνω απ' όλα στην διαπολιτισμική συμβίωση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε μου. Μια πολύ καλή ομιλία. Βέβαια είναι φυσικό η καλύτερη δημοσιογράφος να κάνει μια τόσο πολύ καλή ομιλία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο που μπορέσετε να συμμεριστείτε τι απόψει σα ε, μαζί μα τώρα. Είναι πολύ σημαντικό για μα να ξέρουμε ποια είναι η βάση στην οποία στηρίζεστε και τι πιστεύετε στα... και παρουσιάσετε στα άρθρα σα και βέβαια στο άρθρο που κέρδισε το βραβείο αυτό. Σα ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Περνάμε στην άλλη κατηγορία, στη δεύτερη κατηγορία. Τώρα ο συνάδελφος Πιτέλα είναι εδώ, αντιπρόεδρο, Αυξανόμεθα λοιπόν εδώ. Το επόμενο βραβείο είναι διαδίκτυο, στον τομέα του διαδικτύου. Το βραβείο στην κατηγορία αυτή χορηγείται στον Σλάμ ε, Κομβάλικ από την Ουγγαρία. για το ικανοί καταναλωτές της Βρυξέλλες ε, προχωράνε αυτό παρουσιάζει την Ευρώπη με πολύ καλό τρόπο. Το άρθρο αυτό είναι ιδιαίτερα ανοιχτό και έχει τη δυνατότητα όλο το κοινό να παρεμβεί. Λοιπόν, καταρχήν θα πρέπει να σας το βραβείο. Αυτό για σας. Κυρίες και κύριοι, πριν από μερικές μέρες ήμουνα σε μια ομάδα δημοσιογράφων που ζητούσαν ένα άρθρο που σας προετοιμάζανε για το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, ήμουνα κάπω κάπως σκεπτιστικής. Ε, κάποιος με κοίταξε και είπε μην το κοιτάτε αυτόν. Βέβαια του αρέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του δώσαν ένα βραβείο. Ελπίζω στο μέλλον όταν μιλάω για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Ευρώπη να μην υποσκάπτει το γεγονός ότι έχω το βραβείο την αξιοπιστία μου. Πάντως σας ευχαριστώ πάρα πολύ. δεν έχουμε πολύ χρόνο, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρέπει να προχωρήσουμε τώρα. Λοιπόν, το επόμενο βραβείο για την κατηγορία διαραδιοφωνίας. Ραδιοφωνία. Το βραβείο χορηγείται Ζίγεφ Πρέσνεφ από την Πολωνία για το πρόγραμμα τρίτη φορά ε, τρίτη και καλή τρίτη και καλή ένα πρόγραμμα που αναφέρεται στο δράμα εκείνο των εργαζομένων που απασχολούν στα ναυπηγεία του Στετίνου και προσπαθούν να τηρεί, κρατήσουν την εργασία τους όταν απειλούν τόσες θέσεις απασχόλησης. Συγχαρητήρια. Thank you much. It's uh, you, you probably should take it with you and our colleague. Εδώ το ραβείο για σας. Α, και το, το πρωτότυπο χαρτί ξέχασα να το δώσω προηγουμένω. Θα σας δώσω τώρα το βραβείο σα, αυτό. Κύριε Σμίγεφ Πλέσναρ. Panie jury, i Κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να πω ότι η δική μου εκπομπή ακολούθησε μια προκλητική προσέγγιση. Μίλησα με πολύ επικριτικό τρόπο για την Ένωση και στην εκπομπή μου ακούγονταν και οι φωνέ των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι στρέφονται τουλάχιστον κατά φαινόμενα κατά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πάντω του οποίου πρέπει να ακούσουμε προσοχή, γιατί αυτό που έχω να πω είναι πολύ σημαντικό. Το παράδοξο θα είναι ότι σήμερα εργαζόμενοι άλλων ε, εταιριών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην Πολωνία σήμερα ε, ύψωσαν και αυτή τη φωνή τους για να πούν ότι θα ήθελαν αντίστοιχους όρους της εκαθάρισης ε, για τις εταιρείες τους, όπως ε, αυτούς που ε, επιβλήθηκαν στο ναυπηγείο του Στσένιν. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστώ τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής που εκτίμησαν ε, την εκπομπή μας, τη ραδιοφωνική αυτή εκπομπή, ως γνήσια ραδιοφωνική εκπομπή, γιατί αυτό που φροντίζουμε είναι να μην φαίνεται σαν μία διαφήμιση, αλλά να κάνουμε τη δημοσιογραφία όπως έχουμε μάθει να την επιτελούμε ως λειτουργήμα, πραγματική δημοσιογραφία και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Τζέκος Τσίβας και την κυρία Ποβατόσκα, ε, τους συναδέλφους από το στούντιο της, του ραδιοφωνικού μου σταθμού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν έχω εμπειρία από τέτοιε εκδηλώσει και έτσι δεν ήξερα ότι μπορούσα και να μιλήσω πολωνικά. Βλέπετε, γυράσκω διδασκόμενος. Τα είχα προετοιμάσει όμως όλα τα... ό,τι είχα να πω στα αγγλικά και δεν μπορώ εκ του προχειρού να τα μεταφράσω στη μητρική μου γλώσσα. Την επόμενη κατηγορία λοιπόν τη τηλεόραση και εν τέλει κατηγορία τηλεόραση, το βραβείο δημοσιογραφία απονέμεται στην Έλκε Σάσερ και τον Κρίστιαν Κέλλερ από τη Γερμανία για την εκπομπή ποιος φοβάται την Ευρώπη και πώς ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Πολωνία ντοκιμαντέρ που ε, εστιάζεται πάνω στη ζωή τριών γεωργικών οικογενειών της Πολωνίας ε, μετά την ένταξη της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακολουθεί την καθημερινή του ζωή επί τρία χρόνια και δείχνει πώς επηρεάζεται ο καθημερινός βίος των Πολωνών από την ένταξη και κυρίως των γεωργών. Σας ευχαριστούμε πολύ και συγχαρητήρια. Please και το βραβείο σας. Συγχαρητήρια και σας ακούμε. Λοιπόν, ούτε κέρα είμαι οτι η χρυσές, αλλά απλώς αν το συμβουστώ θα σας πω την ιστορία του, της ταινίας αυτής. Το στην αρχή του 2004 πριν ενταχθούν ε, οι νέε χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε στο γραφείο μα στο Βερολίνο και λέγαμε κάτι πρέπει να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Αυτό που ξέραμε ότι στη χώρα σα, κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν πάρα πολλοί γεωργοί. Και πιστέψαμε ότι η εσωτερική αγορά θα είχε σημαντικέ επιπτώσει στου παραγωγού αυτού. Και σκεφτήκαμε πού να πάμε. Είπαμε να πάμε σε ένα μικρό χωριό κοντά στα χρονικά σύνορα, το λέγεται Κούσινα, και πήγαμε εκεί έτσι, μόνοι, λοιπόν, χωρίς χρηματοδότηση, χωρίς τίποτα άλλο. Και η ιδέα μας ήταν να παρακολουθήσουμε επί τέσσερα χρόνια τι γινόταν στο χωριό αυτό. Βρήκαμε τρεις διαφορετικούς πρωταγωνιστές, όλοι στο ίδιο επίπεδο περίπου. Είχαν μια γελάδα, ένα άλογο, καθένας και ένας με ε, κοστούμι έτσι προσπερβατούσε εκεί στο, στο χωριό αυτό και προσπαθούσε να τους ενημερώσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, είδαμε τι έγινε με τους ανθρώπους αυτούς. Το πρώτο χειμώνα ο Μάτσιν και η Κάσα, ένα ζευγάρι, είχαν χτίσει ένα καινούριο κτίριο και είχαν 100 100 ε, αγελάδες, οι οποίε ήταν Ολλανδικές αγελάδες, illnesses. Που είναι πολύ γάλα. Ένα χρόνο αργότερα, αυτό το ζευγάρι αγόρασε ένα τέος κολχιός στη, στο γοριό αυτό και παίρνανε πάντα ε, βραβείο για τους καλύτερους παραγωγούς. Το μόνο πράγμα ήταν να πάνε και στη Μαγιόργα κάποια φορά, αλλά τα καταφέραν δεν είχαν χρόνο. Ε, ο άλλος Γιώργος δεν άλλαξε τίποτα στη ζωή του. Ξεκίνησε με τρεις αγελάδες και τέλειωσε με τρεις αγελάδες. Και το τρίτο, το τρίτο υπήρχε ε, μια, ένα τραγικό τέλος γιατί την εποχή του κυνηγιού ήταν μεθυσμένος αυτός στο δάσος και τον σκοτώθηκε και πέθανε. Λοιπόν, υπάρχουν κίνδυνοι για όλους, όχι μόνο ευκαιρίες και πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε και την Κριτική Επιστροπή θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μάρτιν Πίπελ που μας έδωσε από την άρτη χρηματοδότηση για να τελειώσουμε το ντοκιμαντέρ αυτό. Σας ευχαριστώ όλους. Λοιπόν, συναδελφοί, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ε, ομιλίες σας, τις πληροφορίες σας, τις εργασίες σας. Σας ευχαριστώ όλους τους εθνικούς ε, νικητές. Ε, οι συνάδελφοι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο πάει εδώ αυξάνονται, βλέπω και πληθύνονται, έρχονται φαίνεται από άλλες συνεδριάσεις. Και όπως σας είπα στην αρχή, δεν μπορούμε να βελτιώσουμε τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε στους πολίτες τι συμβαίνει στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο, στο Λουξεμβούργο, δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τους κάνουμε να πιστεύουν στην πλήρη συμφιλίωση και ολοκλήρωση που χρειάζεται απαραίτητος χωρίς εσάς, χωρίς τους δημοσιογράφους. Σας ευχαριστώ λοιπόν για το θαυμάσιο έργο σας υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για όλους εμάς και για τους πολίτες μας. Σας ευχαριστώ. So we'll make a small pause Ένα μικρό διάλειμμα για πέντε λεπτά και μετά θα συνεχίσουμε με τη συζήτηση των ομάδων. Beach.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

Ladies and gentlemen, good morning. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Έχω διερμηνία στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα ελληνικά, τη δική μου γλώσσα, πολωνικά και γερμανικά. I will speak in Greek. <laughs> Εγώ θα μιλήσω ελληνικά. Ε, καταρχάς, θέλω να σας καλωσορίσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να σας ευχαριστήσω που είσαστε σήμερα μαζί μας σε μια μέρα αφιερωμένη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στους δημοσιογράφους να συγχαρώ με την ευκαιρία τους νικητές του βραβείου δημοσιογραφίας και να ευχαριστήσω επίσης και τους συμμετέχοντες σε αυτό το πάνελ συζήτησης για ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό για την εποχή μας και κυρίως για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι ε, ένα σώμα όχι μόνο νομοθετικό αλλά και ανοιχτό στην κοινωνία. Το θέμα μας λοιπόν σήμερα είναι ο ρόλος των νέων μέσων επικοινωνίας. Μια, είναι μια ευκαιρία για μια δημοκρατία πιο συμμετοχική. Ε, είναι γεγονός ότι Έχουμε όλοι αυτή την προβληματική στη σκέψη μας, το, στη δράση μας, τη σχέση δηλαδή μεταξύ νέων μέσων επικοινωνίας και των παραδοσιακών μέσων επικοινωνίας. Εμείς οι πολιτικοί αναζητούμε να δούμε πόσο τα νέα μέσα επικοινωνίας μας είναι χρήσιμα, πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε, γιατί η τεχνολογία μας δίνει πολλές ευκαιρίες και αναρωτιόμαστε πολλές φορές εάν μπορούμε αυτό το τεράστιο κοινό που μπορούμε να αγγίξουμε με τα νέα μέσα επικοινωνίας, αν είναι συγκεκριμένο, δομημένο, αν μπορεί το μήνυμά μας να φτάσει βαθιά σε αυτούς ή η επικοινωνία μαζί τους είναι επιφανειακή. Απ' την άλλη πλευρά διερωτώμεθα πώς η, τα παραδοσιακά μέσα α, ενημέρωσης, πώς οι δημοσιογράφοι οι ίδιοι ε, αξιοποιούν αυτά τα μέσα επικοινωνίας. Αποτελούν για αυτούς μια πηγή πληροφόρησης, μια πηγή έμπνευσης. Ε, και από την άλλη πλευρά α, διερωτώμεθα πόσο οι δημοσιογράφοι παραδοσιακοί τοποθετούν εμάς τους πολιτικούς στο πλαίσιο αυτής της επικοινωνίας με τα νέα μέσα πληροφόρησης. Ε, αποκαλυπτόμεθα περισσότερο στις πτυχές του πολιτικού μας λόγου, της πολιτικής μας κατεύθυνσης ή απλά εκτίθεται η προσωπική μας ζωή περισσότερο στο κοινό. Είναι ερωτήματα λοιπόν που σίγουρα τα μοιραζόμαστε και η συζήτηση θα αποκαλύψει και πολλά άλλα στη συνέχεια. Θέλω με πολύ χαρά και τιμή να σας παρουσιάσω τους συνομιλητές μας σε αυτό το πάνελ. Εκ δεξιών μου είναι η συνάδελφος και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κυρία Κοχμερίν η οποία είναι και μέλος της ε, ομάδας εργασίας για τα μέσα επικοινωνίας και πληροφόρησης. Έχει και μια ιδιαίτερη επίσης ευθύνη, προεδρεύει του, του, της ομάδας υψηλού επίπεδου για την ισότητα και τη διαφορετικότητα, κάτι πολύ σημαντικό σε σχέση με το θέμα μας, που είναι η δημοκρατική και συμμετοχική κοινωνία. Ε, επίσης θέλω ε, να ε, καλωσορίσω τον κύριο Μόρτεν Λόκετγκάρντ, ε, αντιπρόεδρο της Επιτροπής του Κοινοβουλίου, της Νομοθετικής Επιτροπής, της ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για, την, για τον πολιτισμό, την παιδεία και μέλος της Επιτροπής που εξέλεξε τους σημερινούς νικητές. Είναι επίσης μαζί μας ο κύριος Μίκαλ Στόμπενοφ, από δημοσιογράφος από την εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung, ε, ο οποίος είναι και ειδικευμένο ε, σε θέματα οικονομίας, ε, συνθήκων εργασίας, πολύ σημαντικά θέματα αναδύονται σήμερα πολύ στην επικαιρότητα λόγω της οικονομικής διεθνούς κρίσης και των συνεπειών της σε όλους τους τομείς και τις ομάδες της κοινωνίας μας. Επίσης είναι μαζί μας και η κυρία Λετίτσια Καμπίνη, η οποία είναι μέλος της Επιτροπής ε, του Ευρωπαϊκού Τύπου για την Νεολαία ε, και η οποία έχει μια ιδιαίτερη εμπειρία στις σχέσεις της, ε, της ε, ομάδας αυτής της νεολαίας, της οργάνωσης της νεολαίας με με τον τύπο. Ε, λοιπόν, νομίζω ότι ήδη όλοι έχουμε το ενδιαφέρον να ακούσουμε τους συνομιλητές μας και θα ξεκινήσω από την κυρία Κόχμεριν να δώσω το λόγο. Θα παρακαλέσω τους συνομιλητές... Ε, α, με, ναι, με συγχωρείτε. Ε, ψάχνω μόνο, με συγχωρείτε πάρα πολύ, το πάνελ μας είναι ε, πιο πλούσιο από ό,τι ήδη ανέφερα. Έχουμε μαζί μας, με συγχωρείτε πολύ, και τον κύριο Σλάνκο, ο οποίος είναι ε, δημοσιογράφος από το Ορίγκο Χου, ε, έχει μια ιδιαιτερότητα ε, και θα μας δώσει ενδιαφέροντα στοιχεία διότι έχει εμπειρίες και έξω από την ευρωπαϊκή κοινωνία και από μια ιδιαίτερη χώρα και εγώ την αγαπώ πολύ και ασχολούμαι μαζί της στο Λίβανο που είναι ένα θέατρο γεωστρατηγικών διαφορών και ένα λίκνο καλλιέργειας του συνύπαρξης πολιτισμών και θρησκειών. Ε, περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τη δική σας εισήγηση, κύριε Σλάνκο. Λοιπόν, επανέρχομαι στη συνάδελφο την κυρία Κοχμερίν, θα της δώσω το λόγο. Ήθελα να παρακαλέσω να είναι σύντομες οι παρεμβάσεις, πέντε λεπτών, με ένα κεντρικό στίγμα, όπως όλοι έχετε τη δυνατότητα και την ικανότητα να το κάνετε, για να έχουμε τη δυνατότητα μετά και παρεμβάσεων. Και σας λέω εκ των προτέρων ότι λυπάμαι που θα πρέπει να φύγω 11 παρα 5, γιατί έχω μια άλλη αμετάκλητη υποχρέωση. Ευχαριστώ για την κατανόησή σας. Κυρία Κοχμερίν, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, εξόδημες κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλους. Το θέμα για τη συζήτηση είναι ο ρόλος των νέων μέσων ενημέρωσης. Είναι αυτό μια ευκαιρία και δυνατότητα για περισσότερη δημοκρατική συμμετοχή. Νέα μέσα θα έλεγα είναι ό,τι σχετίζεται με το διαδίκτυο blogs, online ή και η δυνατότητα να δημιουργήσει κανένα μόνο σε ένα πρόγραμμα ταινιών, όλα αυτά μέσα στα πλαίσια των νέων μέσων. Και πάνω σε αυτά θα ήθελα να μιλήσω. Είναι μια δυνατότητα για περισσότερη δημοκρατική συμμετοχή, ναι ή όχι. Θα αρχίσω με ένα πολύ επίκαιρο παράδειγμα που δεν έχει καμία σχέση με πολιτική, αλλά που διευκρινίζει τις δυνατότητες των νέων μέσων. Ορισμένοι από εσάς θα το είδαν ίσως. Η εφημερίδα Frankfurt Allgemeine, μια κλασική αν θέλετε εφημερίδα, το παρουσίασε. Ο Τέικλουμ απέξε το τέταρτο παιδί της. Την ημέρα της γέννησης του παιδιού αυτού ήταν ήδη στα μέσα online. Τέσσερις-πέντε μέρες πριν συμπεριληφθεί στις εφημερίδες. Δεν υπήρχε καμία επίσημη δήλωση ή ανακοίνωση, αλλά στα μέσα online υπήρχαν πολλές ε, εκθέσεις, διάφορα ονόματα για το παιδί, τόπος και ώρα γέννησης. Αναφέρω το. Ορισμένε εφημερίδε και ορισμένε ε, ορισμένες σταθμοί τηλεόραση το πήρανε από τα μέσα αυτά online και το παρουσίασαν. Ορισμένε εφημερίδες και τηλεόρασης περίμεναν όμω να μπορέσουν να το επιβεβαιώσουν, να το ελέγξουν, είναι σωστή η πληροφορία ή όχι. Άρα όταν κάναν την παρουσίαση είχαν κάποιες μέρε καθυστέρηση. βλέπει κανένας ότι υπάρχουν ορισμένες ε, πληροφορίες στα μέσα ε, online πιο ε, νωρίς, αλλά το θέμα είναι, είναι έγκαιρες οι πληροφορίες αυτές, είναι της ε, μορφής με την οποία μπορεί κανένα να εργαστεί, να αποτελέσουν μια βάση ενημέρωσης. Αυτή είναι η δυσκολία που αντιμετωπίζει κανένας γιατί βέβαια το θέμα της ταχύτητας και της επικαιρότητα στήθεται ακόμα πιο έντονα στα νέα μέσα ενημέρωσης. Βρισκόμαστε λοιπόν θα έλεγα σε μια μεταβατική περίοδο όπου οι αρχικές παραδοσιακές μέθοδοι δημοσιογραφίας καλούνται να ερευνήσουν περισσότερο. Στο παρελθόν είχε κανένα τη δυνατότητα να κάνει τι έρευνέ του και να δημιουργήσει μια δική του εικόνα Τώρα υπάρχει ένας αναγωνισμός για μια νέα μορφή καταναλωτών ειδήσεων, αν θέλετε, που δεν ενδιαφέρονται σωστά για τα κλασικά μέσα ενημέρωσης. Τα επόμενα 10-15 χρόνια, φαντάζομαι, θα υπάρχουν τεράστιες αλλαγές. Δεν ξέρω ποιος προς ποια κατεύθυνση. Ούτε εκείνοι που ασχολούνται με το θέμα αυτό το ξέρουν ακριβώς. Ο επικεφαλής του WISE, ένα περιοδικό που ασχολείται ακριβώς με τις εξελίξεις το διαδίκτυο είπε δεν ξέρει προς τα που κινείται η όλη κατάσταση, ξέρει όμως ότι θα υπάρχουν τεράστιες αλλαγές. Αυτό είναι κάτω, κάτι στο οποίο θα πρέπει να προσαρμοστούμε ιδιαίτερα ως πολιτική. Δηλαδή, από τη μια μεριά υπάρχει πιο άμεση, πιο γλίγορη επικοινωνία και υπάρχει και η αναμονή των καταναλωτών να υπάρχουν πιο γρήγορε αντιδράσεις. Από την άλλη μεριά υπάρχει πάντα η υποχρέωση να ελεγχθούν κάποιες ειδήσει και να υπάρξει και μία δυνατότητα περισυλλογής. στο παρελθόν όταν στις εφημερίδες χρειαζόταν μία εβδομάδα για να απαντηθεί μία επιστολή αναγνώστη, η κατάσταση ήταν πολύ διαφορετική. Λοιπόν, πιο γλίγορη, πιο άμεση επικοινωνία, αλλά ο κίνδυνος ότι έτσι παραβλέπεται το γεγονός ότι δεν υπάρχει υποχρέωση να ε, προσπίσει κανένα σε αυτά που έχει πει, που έχει γράψει, με το όνομά του, με την υπογραφή του. Και ο κίνδυνος ότι υπάρχει μια τέτοια πλημμύρα, ένας τέτοιος κατακλυσμός πληροφοριών που δεν μπορεί κανένας πια να τις επεξεργαστεί και να τις κατανοήσει. Εδώ νομίζω θα μπορέσω να διακόψω θα συζητήσουμε τις διάφορες πτυχές των νέων μέσων. Καταρχήν σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ Σιλβάνα. Έδωσε ένα στίγμα πράγματι της δημοκρατικής κοινωνίας και των, α, ε, ομάδων που μπορούν να ενδιαφερθούν και να εμπλακούν. Τώρα θα έχει το λόγο ο κύριος Μόρτεν Λόγκεγκάρντ ο αντιπρόεδρο όπως είπαμε, τη Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίο θα μιλήσει στη μητρική του γλώσσα. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα, βλέπετε εδώ, στα δανεικά. Α, δεν έχουμε. Α, there not interpretation in Danish. Can speak in English? Yes. Yes, yes. Κυρία Πρόεδρε, μπορεί να μιλήσει ε, δανέζικα. Υπάρχει δυνατότητα να μιλήσει δανέζικα ο κύριος. Υπάρχει η δυνατότητα. Υπάρχει. Okay. You can speak Danish. I can speak Danish. Okay. Well, I will do so. Ευχαριστώ πολύ για τη διευκρίνηση της διερμηνής. Well, I thank you very much for for having me here. I'm a I'm a I'm a Dane. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε ασφαλώς ότι είμαι Δανός. Θα συνεχίσω στη μητρική μου γλώσσα γιατί έχουμε διαφορετικές λεπτομέρειες να συζητήσουμε στην συνέχεια και είναι πολύ πιο εύκολο για μένα να μιλήσω δανεικά. Ονομάζομαι λοιπόν Λόκεκαρτ. Με πολύ μεγάλη χαρά έρχομαι εδώ γιατί ήμουν και μέλος της Κριτικής Επιτροπής και οφείλω να πω ότι είμαι σχετικά νέος στην πολιτική. Ένα χρόνο μόνο μετρώ στην πολιτική, αλλά έχω 20 χρόνια εμπειρίας από τη δημοσιογραφία. Και με πολύ μεγάλη χαρά ε, βρίσκομαι σε αυτήν εδώ την Κριτική Επιτροπή από την άλλη πλευρά, αν θέλετε, του, της τραπέζης, ε, δηλαδή εκπροσωπώντας την πολιτική. Εν πάση περιπτώσει όμως δεν μπορούσα και να μην δω τα πράγματα με το μάτι του δημοσιογράφου σε όλη αυτή τη ε, διαδικασία. Πολλά είναι τα κριτήρια τα οποία θα έπρεπε να πληρεί ένας υποψήφιος και μπόρεσα να εξετάσω τα θέματα αυτά υπ' αυτή την οπτική γωνιά. Όπως είπα λοιπόν έχω εμπειρία 20 ετή από την πολιτική δημοσιογραφία, στο πολιτικό ρεπορτάζ στην Δανία θα μπορούσα να σας δώσω κάποια παραδείγματα από τη Δανία για το πώς έχει εξελιχθεί ο τύπος με τα νέα μέσα. Έχουμε λοιπόν τώρα έναν Υπουργό Αμήνης με διάφορα προβλήματα όμως, ε, γιατί κάποιοι από τους υπαλλήλου του, από τους υφισταμένους του, αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν τα νέα μέσα, δηλαδή το ίντερνετ, για να καταγγείλουν ή για να διαμαρτυρηθούν για κάποια προβλήματα που διαπιστώνουν ότι αναπτύσσονται μέσα στο Υπουργείο Αμήνης. Και έτσι δημοσιεύθηκε στα αραβικά ένα κείμενο χωρίς να ζητηθεί η άδεια του Υπουργού από το Υπουργείο Αμήνης. Η κατάσταση λοιπόν είναι δεινή, διότι αυτοί οι υπάλληλοι που χρησιμοποίησαν το ίντερνετ για να δημοσιεύσουν το κείμενο που θέλανε, δεν φαντάστηκαν ότι μπορεί αυτό να απαγορεύεται ή να χρειάζεται προηγούμενη έγκριση. Επίσης βλέπουμε από επιχειρήσεις της Δανίας ότι καταγγέλλονται μέσω των blog, των ιστοημερολογίων ή ιστολογίων, για, επί παραδείγματι, απάτες. Είχαμε μια τεράστια, ένα τεράστιο σκάνδαλο απατών, για το οποίο δεν είχε από ό,τι φαίνεται ιδέα ο γραπτός τύπος της ε, ε, Δανίας, τα οικονομικά φύλλα και από την άλλη αναπτύχθηκε ένας, ε, ε, ένας αγώνας δρόμου για το ιστολόγιο που θα δημοσίευε πρώτο τα σκάνδαλα αυτά, τις απάτες αυτές. Η εν λόγω επιχείρηση της Δανίας προφανώς βρέθηκε πολύ εκτεθειμένη. Άρα βλέπουμε ότι και τα ιστολόγια, τα blog δηλαδή, έχουν πρωτοπόρο ρόλο στην ενημέρωση σήμερα. Θέλω να μιλήσω επίσης για τους δανούς βουλευτές ε, για να σημειώσω ότι χρησιμοποιούμε πολύ το ίντερνετ για την ενημέρωσή μας, αν και τα αποτελέσματα δεν είναι πάντοτε 100% ικανοποιητικά. Ίσως δεν είμαστε όλοι πολιτικοί εν γνώση του γεγονότος ότι χρειάζεται να είμαστε παρόντες στο διαδίκτυο, ότι πρέπει να είμαστε παρόντες στο facebook, να έχουμε ιστολόγιο, να μας δείχνει το MTV, όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά, όπως είπε η Σιλβάνα, δεν πρέπει να λησμονούμε και τι συνέπειες έχουν όλα αυτά. Και έτσι σήμερα βλέπουμε ότι η συμπεριφορά ορισμένων είναι κάπως ερασιτεχνική, σαν τον μαθητευόμενο μάγο, ο οποίος έχει να χρησιμοποιήσει ένα νέο μέσο, το ίντερνετ, χωρίς όμως να ξέρει ακριβώς τι συνέπειες μπορεί να έχει η χρήση του. Νέα μέσα λοιπόν, ναι. Επανάσταση, ναι σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούσαμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέχρι τώρα και ιδιαίτερα όσον αφορά τον τύπο σημαίνει αυτή η τεχνολογική επανάσταση ότι πρέπει ο, ο δημοσιογράφος να επανεφεύρει αυτό, να επανασχεδιάσει το λειτουργήμά του. Πριν από 20-30 χρόνια, πριν εμφανιστεί το ίντερνετ, ξέρουμε ότι η δημοσιογραφία περνούσε μια σοβαρή κρίση ή μη άλλο στην Δυτική Ευρώπη διότι βλέπαμε, επί παραδείγματι, ε, ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα ως προς την προσαρμογή στις νέες συνθήκες γιατί η δημοσιογραφία, πότε σχηματίστηκε ως λειτουργήμα λίγο πολύ στη δεκαετία του 50 διευρύνθηκε, επεκτάθηκε. Με την εμφάνιση λοιπόν του ίντερνετ χρειάστηκε να βρούμε ο καθένας τη θέση του. Φυσικά τα νέα δεν μπορούν ε, να είναι επιπληρωμή, δεν μπορεί να ζητεί κανείς αντίτυπο για να δώσει ενημέρωση, θα πρέπει να είναι δωρεάν ο, ο τύπος, αλλά από την άλλη θα πρέπει να υπάρχει και κάποιος τρόπος να κερδίζουμε χρήματα από την κυκλοφορία, από τη διάδοση μιας είδηση, εφόσον θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο να πληρώνεται ο δημοσιογράφος. Άρα λοιπόν πρέπει να βρεθεί ένας νέος τρόπος για την ε, λειτουργία αυτού του επαγγέλματος θα έλεγα περιμένουμε το, το κετό, δηλαδή το τι θα προκύψει σιγά σιγά ε, ως προς το επάγγελμα αυτό. Βρισκόμαστε στις οδύνες αυτή τη στιγμή και δεν είναι ξεκάθαρο τι μπορώ θα βγει από εδώ. Και δεν ξέρω ακριβώς να σας, να σας προβλέψω ότι πρακτικές συνέπειες θα έχει η εξέλιξη την οποία ζούμε αυτή τη στιγμή για τον δημοσιογράφο και το επαγγελμά του. Όμως μπορώ να διαπιστώσω ότι χρειάζεται σε επίπεδο ευρωπαϊκό να ασχοληθούμε πολύ πιο προσεκτικά με τον τρόπο με τον οποίο ε, καλύπτουμε υπερσυνοριακά προβλήματα, είτε αυτά είναι η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή η σύνταξη, είτε είναι η πάταξη της ε, εγκληματικότητας. Υπερσυνοριακή λοιπόν δημοσιογραφία. Να μια πρώτη πρόκληση. Και ξέρουμε ότι σε επίπεδο Επιτροπής Πολιτισμού έχει αναλυφθεί ένα πρώτο βήμα ε, προσπαθούμε δηλαδή να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση για πιλωτικά προγράμματα για τον λεγόμενο υπερσυνοριακό, για την υπερσυνοριακή δημοσιογραφία. Έτσι δηλαδή ώστε να μπορέσουμε να, ε, να βοηθήσουμε ε, στην ανάπτυξη της ενημέρωσης μεταξύ κρατών όπου υπάρχουν μετακινήσεις πολιτών ή άλλα φαινόμενα ε, υπερσυνοριακά. Αυτό είναι ένα νέο φαινόμενο ε, δημοσιογραφίας που άλλωστε ξέρω ότι προσέλκυσε και την προσοχή μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Θέσατε ενδιαφέροντα ερωτήματα και για εμάς τους πολιτικούς και για τους δημοσιογράφους. Πόσο πρέπει εμείς να ελέγξουμε την ε, ουσία της επικοινωνίας και τη χρήση αυτών των μέσων μαζική ενημέρωση, των καινούριων, τη καινούργια τεχνολογία, αλλά πώ και οι δημοσιογράφοι πρέπει ίσως να επαναπροσδιορίσουν και επανασχεδιάσουν το επάγγελμά τους και το, τον τρόπο λειτουργίας τους. Ε, τώρα το λόγο θα πάρει ο κύριος Σταμπενόβ από την ε, Frankfurter Allgemeine Zeitung ε, για το θέμα α, οπωσδήποτε της οικονομικής κρίσης ε, φαντάζομαι θα αναφερθείτε και το πόσο μπορεί τα νέα μέσα ενημέρωσης να δώσουν ε, πληροφορίε και απαντήσεις στα θέματα αυτά που απασχολούν τους πολίτε είναι το πρώτο ζητούμενο σήμερα από τους Ευρωπαίους πολίτες η αντιμετώπιση της κρίσης και των συνεπειών της. Έχετε το λόγο. Äh, Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλετε νομίζω να σας χαλάσω τη γιορταστική ατμόσφαιρα εδώ αν αρχίσω να σας παρουσιάσω την κατάσταση στα μέσα ενημέρωσης έντυπα και όποια άλλα. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα που μπορούμε να συζητούμε ολόκληρη τη μέρα σήμερα χωρίς να τα λύσουμε. Εγώ θα προσπαθήσω να παρουσιάσω κάτι από σκοπιά ενός ε, δημοσιογράφου στις Βρυξέλλες. Είμαι πολλά χρόνια εδώ. Ε, αντιπρόσωπος για την εφημερίδα Frankfurter Allgemeine. Στην αρχή όταν άρχισα είχαμε τον τηλέτυπο τότε σιγά σιγά ήρθα να γνωρίζω όλα τα άλλα μέσα ε, μέχρι φάξ, ε, μέχρι που φτάσαμε στο, στην εποχή των υπολογιστών που τα πράγματα πάνε τόσο γλίγορα και φτάσαμε στην κατάσταση που γνωρίζετε εσείς όλοι με την έννοια των νέων μέσων εξακολουθώ να έχω προβλήματα. Και εγώ και άλλοι βέβαια. Είναι θέμα ορισμού, γιατί πού είναι η οριοθέτηση. Δεν υπάρχει καμία ε, εφημερίδα, κανένα ραδιοφωνικό ή ε, τηλεοπτικό μέσο ε, ε, εκπομπή που να μην υπάρχει και στο διαδίκτυο. Παραδείγματο χάρη το, το, η εκπομπή, μάλλον το, τα άρθρα του Ζωκα Εμέρ από τις Βρυξέλλες ή του Γιώχ Πίντερ από την Τσάι, του Χάγιο Φρίντριχ, ενός ελεύθερου δημοσιογράφου που έχει ένα μπλοκ που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση Διαφανής διαφανής Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή τα παραδοσιακά μέσα είναι σήμερα τμήμα των νέων μέσων και τα Νάπαλιν ε, σήμερα θα έπρεπε μάλιστα να είναι παρόν ο Ιβτες ο κύριος εκδότης ε, της ε, ε, Βελικής Εφημερίδας The Morgan, όπου είναι παρούσα η εφημερίδα αυτή και και στο διαδίκτυο και <clears throat> ως εφημερίδα. Δηλαδή, ε, έχουμε τη δυνατότητα εργασίας ε, στα νέα μέσα, σύμφωνα με παραδοσιακά, παραδοσιακές αρχές, το, ο παρατηρητής, observer, η parliament που υπάρχει στο διαδίκτυο, που είναι ένα κλασική δημοσιογραφία σε μη κλασικά μέσα στο διαδίκτυο δηλαδή. Εκτός αυτού υπάρχει σαν τμήμα των νέων μέσων αυτών και η δυνατότητα για ε, πολιτικούς δράστες, έχουμε εδώ ορισμένους στο πάνελ, όπου μέσω του διαδικτύου στρέφονται προς την κοινή γνώμη. Είναι αυτό ενδιαφέρον για μας ε, τους δημοσιογράφους, για πρόκειται για πρωτότυπες πηγές ε, Πηγέ της πρώτης γραμμής που μας ενδιαφέρουν εμά τους δημοσιογράφους. Από την άλλη μεριά βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτές οι πηγές έχουν κάποιου πολύ συγκεκριμένου στόχου. Θα πρέπει κανένα πάντα να μπορεί να τι εκτιμά σωστά και με κριτικό πνεύμα. Επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα των blogger των εναλλακτικών ε, δημοσιογράφων επίσης στο διαδίκτυο. Εγώ δεν θέλω να πω ότι όλοι αυτοί είναι ε, άνθρωποι που θέλουν να κάνουν απλώς μια πολεμική χωρίς να είναι κάτι το ουσιαστικό αυτό που έχουν να παρουσιάσουν. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι πάρα πολύ γλίγοροι, ίσως πιο γλίγοροι από την ανάπτυξη της επικαιρότητα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται βάσει διαφορετικών κριτηρίων. Μπορούν να κάνουν πράγματα που εμείς στα παραδοσιακά μέσα δεν μπορούμε να κάνουμε. Θα πρέπει να φροντίσουμε αυτό που γράφουμε να είναι πραγματικά εδρεωμένο, είναι σύμφωνο με την πραγματικότητα και αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία μπορούν να δημιουργήσουν άποψη και γνώμη οι αναγνώστες μας, οι ακροτές μας, οι θεατές μας. Παρ' όλα αυτά συμβάλλουν σημαντικά σε μια μορφή εικόνα των μέσων ενημέρωσης. Παρ' όλα αυτά θέλω και εγώ να συνεχίσω τη δουλειά μου. Πιστεύω ότι εμείς σαν παραδοσιακά μέσα δηλαδή δεν έχουμε παλιώσει τόσο πολύ, δεν είμαστε για πέταγμα θα πρέπει να έχουμε εμείς διαφορετικά κριτήρια, γιατί αυτό που γράφουμε σε εφημερίδες το θεωρούν πολύ ότι είναι πραγματικά αληθές. Κάνουμε μια διάκριση μεταξύ της είδηση και του σχολείου. Τα σχόλια είναι προσωπικά και αυτό θα πρέπει να παραμείνει έτσι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σταμπενόβ. Ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας επισημάνατε για την ε, διαφορετική προσέγγιση, θα έλεγα, την διαφορετική ελευθερία, μορφή ελευθερίας που έχει ο παραδοσιακός δημοσιογράφος από κάποιον που ε, επεμβαίνει, παρεμβαίνει μέσω των νέων τεχνολογιών. Ήθελα να ρωτήσω μήπως ε, πρέπει να δώσουμε τώρα στο ακροατήριο ε, το λόγο, γιατί έχουν ακούσει ε, ενδιαφέρουσες, τρεις ενδιαφέρουσες ε, εισηγήσει, να σχολιάσουμε, να ρωτήσουμε κάτι από αυτόν και να συνεχίσουμε μετά με τους άλλους δύο ομιλητές. Αν συμφωνείτε, να κάνουμε έτσι, να δώσουμε την ευκαιρία στο, στο ακροατήριο να παρέμβει. Ήθελα να ρωτήσω τους παρεμβαίνοντες, να, να τους ζητήσω να είναι πολύ σύντομοι και συγκεκριμένοι, ε, και να παρουσιαστούν ε, ποιον φορέα εκφράζουν και φυσικά το όνομά τους. Λοιπόν, ποιος είναι ο πρώτος που θα πάρει το λόγο. Ο πρώτος ή η πρώτη προσκεκλημένη που θα πάρουν το λόγο. Σας παρακαλώ, έχετε το λόγο. Yes, Yuri from από το περιοδικό Indigo. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι ο δημοσιογράφος μπορεί χάρη στο ίντερνετ να κάνει πιο πολύ έρευνα. Άρα όχι μόνο να παραγάγει, να διαδώσει το έργο του, αλλά και πολύ περισσότερες δυνατότητες να συνεργαστούμε, να βρούμε διεθνείς δυνατότητες συνεργασίας ή νέους συνδεσμούς ή πηγές. Αυτό είναι που δεν ακούστηκε ιδιαίτερα. Αυτό ήθελα να υπογραμμίσω. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Είχα και εγώ αναφερθεί στην ε, σύντομη εισήγησή μου στην αρχή ότι μπορεί να αποτελεί και πηγή πληροφόρησης και έμπνευση το ίντερνετ για τους δημοσιογράφους. Να πάρουμε και τις άλλες παρεμβάσεις και μετά να απαντήσουν ε, οι εισηγητές. Ποιο άλλος θέλει να παρέμβει, να ρωτήσει, να επισημάνει κάτι που χρειάζεται σχολιασμό στη συνέχεια. Με συγχωρείτε, ναι, σας ακούω. Hello, my name is Macarena Rodriguez. I'm... Μαντελένα από την Ισπανία και είμαι ιστολόγος. Θεωρώ αυτήν ιστολόγο, blogger, όχι δημοσιογράφο. Ποτέ δεν δούλεψα ως δημοσιογράφος. Μπορεί να έχω σπουδάσει δημοσιογραφία μένα, αλλά μόνο μέσα από το blog μου έχω δουλέψει. Και αυτό που δεν ακούω αρκετά είναι ακριβώς αυτό, γιατί μιλάτε περισσότερο για το πώς θα πρέπει τα παραδοσιακά μέσα να προσαρμοστούν στα νέα μέσα επικοινωνίας. Αλλά δεν την υπόψη ανθρώπου σαν και εμένα, ανθρώπους που μέσα από το blog, από το Twitter ε, διαδίδουν τις απόψεις τους ε, ή γράφουν μέσα από το Facebook. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τις απόψεις σας και πώς θεωρείτε ότι μπορούν αυτοί οι νέοι άνθρωποι, αυτή η νέα μορφή δουλειάς να ενταχθεί και στα παραδοσιακά μέσα ή αν θα μας αναγνωρίσετε ποτέ ως ισότιμους δημοσιογράφους. Uh, um, Μερικές ερωτήσεις. Είναι ελεύθερος ε, δημοσιογράφος της αναφέρθηκε να υπάρχει ο Μάντοχ λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει πιο πολλή ενημέρωση επιπληρωμή στο διαδίκτυο. Τι λέτε από αυτού, σήμερα η γενιά θεωρεί ότι πρέπει να είναι όλα ελεύθερα στο διαδίκτυο. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή κανένα θα πλήρωνε για τα θέματα αυτά, για τις νέες πληροφορίες για το στο διαδίκτυο ή όχι, αλλά τι άποψη έχετε εσείς και ποια είναι η άποψή σας για το ότι το BBC έχει μια ελεύθερα προσβατή ε, ιστοσελίδα που πληρώνεται από τους ε, φορολογούμενους. Συγκεκριμένη ερώτηση. Άλλη ερώτηση, παρέμβαση. Please. Euh, je suis Aurore Pénois, donc je suis... Euh, Aurore Πενουά, φοιτήτρια δημοσιογραφίας εδώ στις ε, Βρυξέλλες, σπουδάστρια. Είπατε ότι θα πρέπει να είναι δωρεάν η πληροφορία, αλλά δεν είναι λίγο επικίνδυνο να επιμείνει κανείς μια τέτοια ιδέα εάν δεν είναι δυνατόν να πληρωθεί ο δημοσιογράφος, πώς θα κάνει καλά τη δουλειά του. Ωραία. Λοιπόν, δεν βλέπω ενδιαφέρον στη συνέχεια θα μείνουμε εδώ και θα δώσω το λόγο και στους τρεις. Θέλετε όλοι να παρέμβετε, κυρία Αντιπρόεδρε, έχετε να απαντήσετε σε αυτά τα ερωτήματα που θέθηκαν. Ωραία. Η κυρία Κοχμερίν θα απαντήσει πρώτα. Πολύ σύντομα, γιατί και οι άλλοι δύο συνάδελφοι εδώ στο πάνελ θέλουν να πάρουν το λόγο σίγουρα. Καταρχήν θεωρώ ότι για τους πολιτικούς, όπως ακούσαμε και προηγουμένως, η σημασία των blogs και των Twitter στην Ευρώπη είναι διαφορετική από ότι ίσως στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Άμα δούμε τις ευρωεκλογέ, δεν θέλω να θεωρηθώ κοινική, αλλά κοιτάξτε, ποιοι πάνε να ψηφίσουν στη Γερμανία είχαμε κάτι παραπάνω από το 40% συμμετοχή στις εκλογές. Και 70% αυτών των ανθρώπων ήταν πάνω από το 65%. Εγώ γράφω blog, τακτικά. Έχω σελίδα στο facebook, στο neutral κλπ. Αλλά δεν φτάνω στους εκλογείς έτσι. Πάρα πολύ λίγο. Ως πολιτικός δηλαδή θα πρέπει πάντα να σκεφτώ πριν από τι εκλογέ πώ θα φτάσω να αγγίξω εκείνου τον οποίο την ψήφο επιθυμώ. Είναι τώρα νομίζω μια μεταβατική κατάσταση. Θα αλλάξω τα πράγματα με τι εξελίξει δημογραφικέ. Αυτό που αναπτύσσεται δυναμικά, blog, twitter και ό,τι άλλο υπάρχει, από σκοπιάς πολιτικών δεν είναι επαρκές γιατί δεν φτάνει στους απαραίτητους εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπορεί να υπάρχει μια εξέλιξη στο μέλλον. Και να μπορεί να περάσει από εκεί βέβαια στα μέσα τα οποία καταναλώνουν περισσότερο οι εκλογές. Αν δούμε τι γίνεται σε άλλα μέρη του κόσμου, τι επανάσταση έλαβε χώρα με τη δυνατότητα αυτή των ΜΜΕ με τις νέες ε, επικοινωνίες, παραδείγματος χάρη κάτι άλλο, κινητή τηλεφωνία. Υπάρχει παντού σε όλο τον κόσμο πολύ περισσότερα δεδομένη από ό,τι έντυπα μέσα. Μπορεί κανένας μέσω του κινητού του τηλεφώνου να πάρει επίσης πληροφορίες. Και έτσι σε μια περιοχή στην οποία δεν υπάρχουν τόσες πολλές πληροφορίες, γιατί δεν υπάρχει ο γραπτός τύπος κλπ. Υπάρχει δυνατότητα να συμμετάσχουν και οι άνθρωποι αυτοί μέσα των κινητών τους τηλεφώνων. Αλλά αυτό αλλάζει πολύ για τον διαβάσει κανένα μια εφημερίδα. Σημαίνει ότι ίσως αρχικά ενδιαφέρεται για ένα άρθρο, παίρνει την εφημερίδα και μετά διαβάζει και κάποιο άλλο τομεί και διαβάζει περισσότερα από εκείνα που διάβαζε, θεώρησε στην αρχή ότι θα το ενδιαφέρουν. Ενώ τώρα μπορεί κανένα να συγκεντρωθεί σε αυτό που εκ μια αρχής τον ενδιαφέρε. Η επιλογή δηλαδή ε, του τι διαβάζει, τι κοιτάει κανένας, περιορίζεται έτσι. Τώρα δεν ξέρω καλό, κακό, δεν έχω να πω και η δυνατότητα ορισμένων ε, μέσων ενημέρωσης μόνο περιορίζεται. Τώρα το θέμα της εκπαίδευσης των δημοσιογράφων. Ναι, παλιά η εργασία των πολιτικών, παραδείγματος χάνει, χρειάζεται να περάσει μέσω των ε, αρχείων της εφημερίδας ή της βιβλιοθήκης για να μπορέσει ο δημοσιογράφος να έχει τις πληροφορίες αυτές, τώρα στο διαδίκτυο βρίσκει τα πάντα. Και ξέρουμε ότι εκείνοι που γράφουν στο ε, facebook για το τι έκανα στο τελευταίο πάρτι ίσως τα βρουν μπροστά τους όταν ο επόμενος εργοδότης κάτσει και διαβάσει και προσπαθεί έτσι να γνωρίσει τον υποψήφιο. Αλλάζει η κοινωνία σημαντικά. Ο κύριος Λόκιγκορντ έχει το λόγο. Øh, Ευχαριστώ πολύ. Πολλές ε, ερωτήσεις, ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Η πρώτη αφορούσε την ε, δωρεάν παροχή της ενημέρωσης. Όχι, εγώ δεν είπα ότι πρέπει να είναι δωρεάν η ενημέρωση. Εγώ είπα ότι είναι σήμερα δωρεάν η ενημέρωση, η πληροφορία δηλαδή σε πολλά από τα ε, site, από τις ιστοσελίδες στο ίντερνετ. Και αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο πρέπει να δεχθούμε. Δηλαδή είναι δωρεάν η ενημέρωση στο ίντερνετ. Πώς θα επιβιώσουμε εμείς που μέχρι τώρα πληρωνόμασταν. Δεν είπα λοιπόν ότι πρέπει να μείνει δωρεάν. Είπα ότι είναι δωρεάν και πρέπει αυτό κάπως να το εξετάσουμε. Βάσει αυτού του χαρακτηριστικού του δωρεάν να προχωρήσουμε. Εγώ, φιλελεύθερος πολιτικά, θεωρώ ότι οι δυνάμεις της αγοράς ρυθμίζουν ε, τα ζητήματα μόνες τους. Στην περίπτωση της δημοσιογραφίας, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είμαι λιγότερο φιλελεύθερος. Και είμαι πεπισμένος ότι η δημοσιογραφία, η ποιοτική δημοσιογραφία εννοώ, ε, ε, για να επιβιώσει σε τον σύγχρονο κόσμο πρέπει να επαναδιατύπωθεί, να επανασχεδιαστεί. Και πρέπει να δούμε τι σημαίνει δημόσια δημοσιογραφία, τι σημαίνει κρατική δημοσιογραφία, σε ποιο βαθμό δηλαδή οι κρατικές αρχές θα επιτρέψουν την ελευθερή ε, ε, διεργασία, την, ελεύθερη ε, λειτουργία της δημοσιογραφίας χωρίς παρεμβάσεις και χωρίς να θέλω να προσβάλλω ή να ενοχλήσω τους Ιταλούς συναδέλφους βλέπουμε στη χώρα αυτή ότι δημοσιογραφία βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση, σε αδιέξοδο θα έλεγα, γιατί μερικές φορές μπερδεύεται, συχαίεται η έννοια του πολιτικού και των μέσων μαζικής ενημέρωσης και άρα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις πολιτικές στην υπόθεση αυτή. Πολιτικά λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει το πόσο θα μείνουν και ανεξάρτητα και ασφαλή τα μέσα αλλά και πώς θα χρηματοδοτούνται. Εμείς στη Δανία έχουμε παραδόσεις για τις οποίες αισθανόμαστε ιδιαίτερη παρήφανοι. Εγώ, παραδείγματι, επί 15 χρόνια εργάστηκα στον κρατικό σταθμό της Δανίας, στο δεύτερο μεγαλύτερο σταθμό, τηλεοπτικό σταθμό της χώρας. Έχουμε δύο ε, τηλεοπτικούς σταθμούς, οι οποίοι ε, απορροφούν το 80% της τηλεθέασης. Αυτό σημαίνει ότι ε, εγγυούμαστε μια ποιοτική δημοσιογραφία. Φυσικά, για να εξασφαλιστεί αυτό, το κράτος επιδοτεί τους σταθμούς. Και άρα νομίζω ότι αυτός είναι ένας τρόπος να προχωρήσουμε. Ε, γι' αυτό, όπως είπα, δεν είμαι τόσο φιλελεύθερος στις απόψεις μου όσον αφορά τη δημοσιογραφία. για την έρευνα που είπατε κάποιος άλλος από την αίθουσα ότι διευκολύνει το ίντερνετ. Όντως, όντως, ποτέ δεν είχαμε τόση δυνατότητα για έρευνα, για διερεύνηση μιας υπόθεσης. Αλλά δεν είναι εδώ το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ο διάβλος διάδοσης της ενημέρωσης. Αυτό που είπε και ο συνάδελφος νωρίτερα. Ναι, τεχνολογία έχουμε. Τηλεοπτικούς σταθμούς έχουμε. Αλλά πόσο τα χειριζόμαστε όλα αυτά. Μας κατακλείει αυτή η πληθώρα πληροφοριών και πρέπει να επιλέξουμε αυτό το οποίο θα διαδώσουμε εμείς, αυτό που θα εκπέμψουμε εμείς αν θέλετε, πώς θα φτάσει στον πολίτη. Το πρόβλημα είναι η κυκλοφορία, η διανομή της πληροφορίας, της ενημέρωσης. Και ποιος θα είναι ο υπεύθυνος για αυτή την κυκλοφορία της πληροφορίας, ποιος θα είναι ο εγγυητής του ότι ο φύχηψη σταθμός δεν θα πέσει στα χέρια κάποιου ο οποίος θέλει απλώς να ελέγξει την αγορά, την πολιτική, το κοινό. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει με κάποιο τρόπο να ρυθμιστούν. Έχουμε να κάνουμε με μεγάλες δυνατότητες που όμως πρέπει να διοχετευθούν κάπως για το μέλλον. Όντως, η έρευνα προσφέρεται άπειρες ευκαιρίες για έρευνα ανά τον κόσμο. Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε και τους διάβλους της διάδοσης πληροφορίας. Υπάρχει η διαφήμιση επίσης. Επίσης υπάρχει και το ζήτημα της σύνταξης της ε, πληροφορίας και επικοινωνίας. Θα ήθελα να πω ότι όταν μιλάει ο κύριος Λόκικαρτ εδώ για κρατικά μέσα, ε, δεν μιλάμε για νέα μέσα, αλλά μάλλον για τα παλαιότερα των μέσων ενημέρωσης και που πρέπει και αυτά να διατηρήσουν τις θέσεις τους για να εξασφαλίζεται η ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Ξέρουμε ότι δεν είναι ανεξάρτητη η δημοσιογραφία των κρατικών μέσων μαζικής ενημέρωσης στο βαθμό που είναι ανεξάρτητη στα, στους κρατικούς σταθμούς της Δανίας, δεν είναι σε όλα τα κράτη έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα πρέπει και να υποτιμούμε το γεγονό ότι από το ίντερνετ, ναι, μεν προσφέρονται πολλέ δυνατότητε, είναι χρήσιμο το ίντερνετ για όλου. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα που αναφέρατε κι εσεί για τη συνεργασία πέραν των συνόρων διαφόρων ειδών μέσων μαζικής ενημέρωσης, διεθνώς ακόμη. Πολύ ωραία όλα αυτά τα αξιοποιούμε όλοι και πρέπει να τα αξιοποιούμε. Αλλά εδώ έρχεται το ερώτημα σε ποιο βαθμό μπορούν τα νέα μέσα να αποτελέσουν τμήμα των παραδοσιακών μέσων ή αν θέλετε που βρίσκεται η διαχωριστική γραμμή μεταξύ παλαιών και σύγχρονων μέσων. Αυτό που ρώτησε η συνάδελφος νωρίτερα. Υπάρχουν μέσα σύγχρονα τα οποία ακολουθούν τις παραδοσιακές δημοσιογραφικές δυνα... Ε, μεθόδους. Αλλά βέβαια οι bloggers, ε, ιστολόγοι έχουν ίσως κάπως πιο αυθόρμητο τρόπο εργασίας. Δεν είναι τόσο παραδοσιακή η οι μεθ... παραδοσιακές μέθοδες, μέθοδοι που χρησιμοποιούν. Αυτό είναι και ένας λόγος για τον οποίο θεωρώ αιτιολογημένη μια κάποια επιφυλακτικότητα έναντι των ε, νέων αυτών μέσων. Επίσης έγινε λόγος ε, για την ε, πρόθεση του Ρούμπερτ Μέρντοχ να ζητήσει μέσω του ίντερνετ πληρωμή για την ε, πληροφορία που διαδίδεται. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει. Όπως είπε ο συνάδελφος, η ανταγωνιστικότητα θα είναι ίσως ο καταλυτικός παράγοντας, το κατά πόσον δηλαδή θα υπάρχει κάποιος άλλος ανταγωνιστής ο οποίος θα προσφέρει την ίδια πληροφορία, επιπληρωμή ή μη. Από εκεί θα κρυφθούν όλα αυτά. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει πληρωμή. Αυτά νομίζω πρέπει να τα πούμε ξεκάθαρα. Και τους εισηγητές και τους προσκεκλημένους μας για αυτόν τον ενδιαφέροντα διάλογο. Ήδη αναδεικνύονται οι πτυχές διαστάσεις αυτής της σχέσης μεταξύ παραδοσιακών και νέων μέσων ενημέρωσης και τη σχέση που έχει η πληροφόρηση και για τους πολιτικούς και για τους δημοσιογράφους και για την αγορά. Ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο κύκλο παρεμβάσεων. Θα πάρει το λόγο ο κύριος Μπάλιντ Λάνκο από την Ουγγαρία, όπως σας είπα. Έχετε το λόγο. Θα ήθελα να εξετάσω το θέμα που έθιξε ο συνάδελφος εκεί. Κατά... Ε, είμαι υπέρ του να, υπάρχουν, να υπάρχει πληρωμή για τα νέα. Εγώ δεν πίστευα ποτέ ότι θα πρέπει τα... <clears throat> οι πληροφορίες να είναι δωρεάν. Δεν το πίστευα ποτέ αυτό. γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ανταποκριτές παραδείγματος χάνει σε περιοχές ε, εμπόλεμες είναι πανάκριβοι. Δεν μπορεί να είναι δωρεάν όλα αυτά. Είναι καλό κάποιος να πληρώνει. Δεν ξέρω κατά πόσο θα λειτουργήσει το σύστημα. Υπάρχουν βέβαια πληροφορίες, ε, ε, ε εφημερίδες που βασίζονται μόνο στις διαφημίσεις και κερδίζουν αρκετά. Οι περισσότερες όμως ξέρω ότι έχουν οικονομικά προβλήματα ακριβώς γιατί χάνουν τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο, στο θέμα όπως το Google News παραδείγματος χάρη και θα πρέπει να υπάρχει κάποιο νέο σύστημα για να πληρωθούν. Και γι' αυτό θα πρέπει κανένα να αποδεχθεί ότι οι ειδήσει οτιδήποτε άλλο πρέπει να πληρώνονται. On your point about, about paid for κατά πόσο θα πρέπει να πληρώνει για τι ειδήσει τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, Καταλαβαίνω που λέτε, πολλοί δεν θα ενδιαφέρονται. Υπάρχουν αρκετοί όμω νομίζω που θα ενδιαφέρονται αρκετά για να πληρώσουν. Εγώ τέσσερα-πέντε χρόνια εργαζόμουν για μια τέτοια ειδησιογραφική εταιρεία και ήταν εντάξει νομίζω. Δεν κερδίζαμε πάρα πολλά, αλλά οπωσδήποτε μπορούσαμε να διατηρηθούμε. Ευχαριστώ πολύ για τη συγκεκριμένη τοποθέτησή σας. Η κυρία Καμπίνη τώρα έχει το λόγο να δούμε πώς βλέπει η νέα γενιά που είναι η γενιά της νέας τεχνολογίας και των νέων μέσων ενημέρωσης. Thank you <clears throat> very much. Um, as first, when I read the title of the panel, I was very interested in seeing that there is uh, three different things. Υπάρχουν ε, τρία διαφορετικά πράγματα που ενδιαφέρουν. Καταρχήν το θέμα της έκφρασης, η έκφραση νέα μέσα. Δεν ορίζεται αυτό στην εργασία μας. Τι είναι το νέο μέσο, τι είναι το παλιό μέσο. Το δεύτερο, η δημοκρατική συμμετοχή. Είναι κάτι που θα πρέπει επίση να οριστεί στον τίτλο αυτού του σεμιναρίου. Χωρίς να περάσω τώρα σε φιλοσοφική συζήτηση βέβαια, νομίζω ότι τα μέσα του Web 2.0 που είναι ο δικός μου ορισμός για το, τα νέα μέσα είναι στην καθημερινή μας ζωή, τα Twitter, το Facebook κλπ. Αυτό είναι κάτι που ξέρετε όλοι νομίζω και σκέφτομαι ποιοι είναι οι χρήστες αυτής της τεχνολογίας. Οι χρήστες της τεχνολογίας στατιστικά είναι οι νέοι διάβαζα ένα άρθρο για, το για την ελεύθερη ιστοσελίδα του BBC που έλεγε ότι 75% των νέων μεταξύ 16 και 24 δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς το διαδίκτυο. I'm 25 right now. Um, Εγώ είμαι πάνω από το όριο αυτό τη ηλικία και ομολογώ ότι θα μπορούσα να ζήσω χωρί διαδίκτυο, κατά πάσα πιθανότητα. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ τι αλλαγέ που θα εισέρχονται στη ζωή μου χωρί το διαδίκτυο. Και η εργασία μου βέβαια ω δημοσιογράφου δεν μπορώ να φανταστώ. Ο κύριος ε, Στάβενοφ θυμάται όταν εργαζόταν με μολύβι και με τηλέτυπο, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ πως δεν εργαστήκα ποτέ χωρίς υπολογιστή. Σήμερα το πρωί δεν μπορούσα να τυπώσω και έπρεπε να γράψω σημειώσεις μου και ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα που δεν μπορούσα να αντιγράψω ε, τα κομμάτια του κειμένου μέσα στο, ε, στην ισοσελίδα μου. Καταλαβαίνω, η κυρία να αναφέρθηκε σε μια μεταβατική περίοδο. Η μεταβατική περίοδος αυτή όμως νομίζω ότι κάποια στιγμή θα φτάξει στην κατάληξή της και τότε όχι μόνο θα έχουμε υιοθετήσει τις νέες τεχνολογίες, αλλά οι νέες τεχνολογίες θα είναι τα πραγματικά μέσα για επαγγελματική δημοσιογραφία και για τον συσχετισμό μεταξύ των δημοσιογράφων, των πολιτών και των πολιτικών. Νομίζω ότι οι στόχοι του Twitter, των blogs και των νέων μέσων είναι διαφορετικοί ίσως ε, από εκείνους των ε, ε, bloggers που είναι πάνω από τα 64, αλλά δεν έχει σχέση αυτό με το γεγονός ότι δεν πάνε να ψηφίσουν οι νέοι, ίσως γιατί δεν τους έχουν πείσει οι πολιτικοί. Νομίζω ο ρόλος της δημοσιογραφίας σήμερα είναι ταυτόχρονα να είναι πιο γλυγόρη και πιο ε, αλληλένδετη και ίσως πιο αναφερόμενοι καλύτερα στην ε, επικαιρότητα και μπορεί να μεταβιβάζει λογικά μηνύματα, σημαντικά μηνύματα. Παραδείγματος χάρη εδώ έχουμε ένα δίκτυο νέων δημοσιογράφων στην Ευρώπη Γιατί αυτό που είναι σημαντικό σήμερα είναι να έχουμε ευρωπαϊκή δημοσιογραφία και αν κοιτάξετε εδώ βλέπετε ότι είναι πολλοί νέοι εδώ. Υπάρχουν 40 νέοι δημοσιογράφοι, νεαροί δημοσιογράφοι που έφερε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ σε αυτό το όργανο που είναι όπως είπαμε προηγουμένως η καρδιά της Ευρώπης τους έφερε εδώ για να δείξει ότι είναι δυνατόν κανείς να παρουσιάσει την Ευρώπη όπως πρέπει. Ίσως είναι ανοιχτά διαδέσιμες οι ειδήσει αυτές στο διαδίκτυο, ίσως πληρώνονται. The profession to be... Ίσως ε, θα μπορέσετε όμως έτσι να όντας η νέα γενιά των δημοσιογράφων να χρησιμοποιήσετε τις νέες τεχνολογίες και να βοηθήσετε τους ε, Ευρωπαίους πολίτες περισσότερο από ό,τι μπορεί να γίνει αυτό. ποτέ. αυτό λείπει νομίζω από τη συζήτηση. Το τι μας βοηθούν να κάνουμε οι νέες ε, τεχνολογίες είναι να έχουμε ευρωπαϊκή δημοσιογραφία. Να μπορούν οι ειδήσει μας να είναι διαθέσιμες σε όλους παντού στην Ευρώπη ταυτόχρονα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που υπάρχει. Και τα προβλήματα που υπάρχουν ε, ξεπερνούνται ίσως με το διαδίκτυο, γιατί αν έχει κανένας ε, ε, έναν υπολογιστή μπορεί να έχει τις ειδήσει σε πολλές γλώσσες ε, από πολλές χώρες και αυτό θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρωτότυπα, δημιουργικά, για να υπάρχει πραγματικά νέα δημοσιογραφία που κατά τη γνώμη μου είναι η ευρωπαϊκή δημοσιογραφία. I the new media. Μάλιστα σε σχέση με τα νέα μέσα του τύπου το καινούριο είναι ότι μπορεί να υπάρχει η κριτική, ας το πω έτσι, έκφραση, διότι χάνουμε ε, την ε, αίσθηση των ε, φρουρών των πυλώνων. Έχουμε λοιπόν πρόσβαση σε αυτό και κάθε ένας φυσικά έχει το καθήκον να κάνει μια επιλογή και μια σχετική σκόπιμη επιλογή. Αυτό όμως επιτρέπει να ακουστούν οι ε, κριτικές φωνές που δεν ήταν πάντα διαθέσιμες στο παρελθόν. Και αυτό είναι εκείνο το οποίο χαρακτηρίζει τον ανεξάρτητο χαρακτήρα των δημοσιογράφων, της δημοσιογραφίας. Εγώ είμαι Ιταλίδα, παίρνω τα σχόλια όπως και πιο πριν το σχόλιο του ότι δεν είναι τόσο εύκολο να υπάρχει ελεύθερη δημοσιογραφία σήμερα στη χώρα μου στην Ιταλία. Και θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα ανάγλυφο παράδειγμα. Το πραγματικό παράδειγμα εδώ μπορεί να υπάρξει ένας νέος ελεύθερος χαρακτήρας της δημοσιογραφίας στα νέα μέσα του τύπου. Να προβληματιστείτε γι' αυτό, όχι να προσαρμοστείτε, αλλά να δημιουργήσετε μια νέα μορφή, ένα νέο είδος ανάπτυξη του επαγγέλματος του δημοσιογράφου. Ευχαριστώ. And just to conclude, <laughs> sorry. Να ολοκληρώσω δύο λόγια ακόμα και ολοκληρώνω. Θα ήθελα να σας πω ότι Κουράστηκα πια να ακούω ότι η ΕΠΑ είναι τόσο προηγμένες στα νέα μέσα του τύπου. Δεν με ενδιαφέρει αυτό, δεν με ενδιαφέρει. Εμείς εδώ στην Ευρώπη είμαστε διαφορετικοί. Είμαι υπερήφανη γι' αυτό και είναι το μόνο που θα ήθελα να αναφέρω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Καμπίνη για την παρέμβασή σας. Ε, πραγματικά δώσατε μια νέα διάσταση στη συζήτησή μας, ε, τη θέση που έχει η δημοσιογραφία σε σχέση με τις ευρωπαϊκές ειδήσει, τις ειδήσει των Βρυξελών δηλαδή και την απήχησή τους στη ζωή των πολιτών, στον, ε, εθνική πολιτική. Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον για μας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι έχουμε μια ολόκληρη πολιτική, ε, πολύπτυχη, γύρω από την επικοινωνία. Ε, οι στατιστικές είναι θαρρυντικές. Ε, όλο και περισσότεροι πολίτες παίρνουν το μήνυμά μας, ακόμη και το μήνυμα της ευρωπαϊκής καμπάνιας, της θεσμικής καμπάνιας που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις ευρωεκλογές. Βέβαια, ένα άλλο θέμα έθεσε η κυρία Κοχμερίν, πώς πείθουμε τους Ευρωπαίους πολίτες να πάνε να ψηφίσουν. Αυτό είναι μια άλλη παράμετρο στην οποία εξετάζουμε και η οποία δεν απαντιέται εύκολα γιατί επισέρχονται πολλά θέματα εκεί, όχι μόνο η απήχηση της καμπάνιας και της επικοινωνίας μας, αλλά και πόσο επηρεάζει την πρόθεση ψήφου η, εθνική πολιτική κατάσταση σε κάθε χώρα. Είναι ένα θέμα το οποίο σας απασχολεί και μας απασχολεί και εμάς, αλλά είναι σημαντικό ότι η κυρία Καμπίνη έθεσε πράγματι το θέμα της ε, δημοσιογραφίας για την ευρωπαϊκή πολιτική, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ανοίξουμε τη συζήτηση με τους προσκεκλημένους μας, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Ζλάνκο, διότι στην ε, πρωτολογία του αφιερώθηκε στο να απαντήσει σε ε, ερεθίσματα που ήδη υπήρχαν από το κοινό και δεν έκανε μια γενική τοποθέτηση. Έχετε λοιπόν το λόγο τώρα να κάνετε μια σύντομη γενική τοποθέτηση. Αν μας αναφερθείτε κι εσείς στο στην ευρωπαϊκή δημοσιογραφία, την, Ευρω... Ε, δημοσιογραφία για τα ευρωπαϊκά θέματα θα είναι πολύ σημαντικό. Έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομε ε, λίγε κάποιε παρατηρήσει, και χωρί να ακούσω το ε, το χρησιμοποιώντας τον, την νέα δημοσιογραφία για τον, τα νέα μέσα του τύπου έχουμε πολλά blogs και δεν είναι όλα αυτά δυνατόν να ενταχθούν στο Twitter, στο ή ε, στο YouTube, αλλά η κύρια συνεισφορά είναι οι καλά ενημερωμένοι πολίτες και δεν είναι τόσο προφανές για μένα ότι όλο και περισσότερο οι πιο σαφείς ε, τοποθετήσεις και εκφράσεις θα συνεισφέρουν υποχρεωτικά σε αυτό. Μία από τις συνεισφορές των νέων μέσων του τύπου στα τελευταία χρόνια ήταν να υπάρξει ο πληθυσμό εκείνων των ε, μέσων που παρήγαν υψηλού επίπεδου ε, πληροφορίες. Θα είναι πολύ δύσκολο να βρείτε τέτοιου είδου ε, δημοσιογράφου υψηλή ποιότητα για τα εξωτερικά θέματα ή στα blogs διότι δεν ε, εισπράττουν χρήματα, δεν βγάζουν χρήματα εκεί και όλα αυτά κοστίζουν πάρα, πολύ χρήματα, πάρα πολλά χρήματα. Και έτσι έχουμε εδώ και την παλαιομοδίτικη αυτή πτυχή των παλαιών μέσων ενημέρωσης όσον αφορά αυτού του είδους την έκφραση και πάλι εδώ θα πρέπει να εστιαστούμε, να υπογραμμίσουμε περισσότερο την ποιότητα του περιεχομένου και όχι τόσο την πλατφόρμα ή το μέσο με το οποίο παρέχεται μια πληροφορία. Ε, πάνω στο οποίο βλέπουμε ότι σε αυτό εδράζεται και οικοδομείται η θεωρία των νέων μέσων. Και όσον αφορά την, τα θέματα της δημοκρατίας, ε, όλο και περισσότερες φωνές ε, έλεγε κανείς ότι θα ενημερώνουν και θα βοηθούν μια καλύτερη συζήτηση και θα αναβαθμίζουν το τελικό αποτέλεσμα. Και πρέπει να δούμε κατά πόσο αληθεύει αυτό και ότι θα καταφέρουν στο τέλος αυτά να βοηθήσουν να λύσουμε κάποια θέματα με εσωτερικού είδους ε, έκφραση των πολιτών ε, τύπου ε, δημοψηφισμάτων όπως αυτά τα θέματα που μπορεί να τίθενται στο ίντερνετ. Είναι ένα εργαλείο, ένα μέσο που πρέπει ιδιαίτερα προσεκτικά να αντιμετωπίσουμε. Δεν είμαι πεισμένος ότι μπορούν με τέτοιου είδους ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα να ρυθμίζονται τέτοια θέματα και δεν θα έπρεπε καθόλου να τίθενται σε δημοψηφίσματα διεθνεί συνθήκε ή σύμφωνίε. Δεν είμαι καθόλου βέβαιο αν με αυτόν τον τρόπο συνεισφέρουμε αν συζητώντας τόσο περίπλοκα σύνθετα θέματα μπορεί να στεφτεί με επιτυχία το εγχείρημα σε ένα τέτοιου είδους δημόσιο ε, ας το πω έτσι ε, φόρουμ όπως αυτά τα δημοψηφίσματα στο ίντερνετ. Όσον αφορά τα θέματα της πολιτικής ε, και τα νέα μέσα του τύπου το χαρακτηριστικό είναι η απουσία ηγεσία σήμερα κυριότερα και όχι η απουσία έκφρασης ή η έλλειψη διαφορετικών φωνών στο φάσμα που εκφράζονται και την ιστορία με τον Winston Churchill που του είχαν πει ότι θα έπρεπε να ακούει πολύ καλά τι λένε οι πολίτες, να ακούει περισσότερο ποια είναι η άποψη των πολιτών. Και είπε ότι οι ε, Βρετανοί πολίτες δεν σεβόντουσαν κάποιο πολιτικό που θα ακολουθούσε μια τέτοια προσέγγιση. Και εδώ λοιπόν αυτό είναι το θέμα σε σχέση με την πολυφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και ενδιαφέρουσε απόψεις. Και τώρα ο λόγο σε εσά. Ποιο θέλει να παρέμβει. Ήδη έχουμε το πρώτο αίτημα. Σα ακούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, είναι δύσκολο να συμφωνήσω με αυτή τη διάκριση νέων και παλιών ε, μέσων. Ε, εγώ άρχισα να εργάζομαι πριν από 30 χρόνια ως δημοσιογράφος. Τότε είχαμε ε, μαγνητοτενίες, μετά περάσαμε στα ψηφιακά μέσα, στο διαδίκτυο και η μόνη διακρίση που μπορούμε να κάνουμε είναι καλή ή κακή δημοσιογραφία. Είτε μεγάλο είναι καλή στην ηλικία, είτε νέο και ποια τεχνολογία χρησιμοποιεί, είναι δευτερεύουσα σημασία. Για μένα το διαδίκτυο είναι ένα θαυμάσιο μέσο καταπληκτικό που επιτρέπει να ζήσουν περισσότερο τα, οι εργασίες μου, οι παραγωγές μου. Δεν περνάνε απλώς από την ε, τηλεόραση και φεύγουν. Αν κάποιος ακούσει κάτι λίγο στο ραδιόφωνο και θέλει μετά να ακούσει το υπόλοιπο, μπορεί να το βρει στο διαδίκτυο υπάρχει συνεχής αλλαγή, συνεχής πρόοδος, βελτιώνουμε την εργασία μας, χρησιμοποιούμε τις τεχνολογίες και αυτές οι τεχνολογίες, εάν μπορούν να κάνουν την εργασία μας καλύτερα ή πιο ευνόητη ή εάν αυτό που κάνουμε βοηθάει τον ακροατή, τον αναγνώστη και τις ίδιες τις ιδέες καλύτερα, αυτό είναι νομίζω μια πολύ θετική εξέλιξη θα είμαστε όλοι ευτυχείς να έχουμε νέα καλά μέσα στα χέρια μας, εργαλεία στα μέσα μας. Μπορούμε έτσι να είμαστε πιο γλίγοροι και με περισσότερη βάση. Πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση της ε, διαχρονικότητας και της ποιότητας που εξασφαλίζουν οι νέες τεχνολογίες. Άλλος παρεμβαίνων. Please. Uh, hello, uh, my name is Stephen Carroll. I'm here εκπροσωπώ την ε, Εθνική Ιρλανδική Ραδιοφωνία και θα ήθελα σε σχέση με την παράδοση για την διεξαγωγή δημοψηφισμάτων. Νομίζω είναι καλή ιδέα αυτή και σίγουρα ζω τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και βλέπω τη συζήτηση αν θα υπάρξει λέει δημοψήφισμα ή όχι για την ε, συμμετοχή και ολοκλήρωση στην Ευρώπη. Και αυτό είναι πολύ καλό και το ενδιαφέρον είναι σε σχέση με τα, την εκστρατεία για το δημοψήφισμα για την συνθήκη της Λισαβόνα στην Ιρλανδία είναι ότι τα κοινωνικά μέσα, δηλαδή η κάλυψη του κενού που υπήρχε και παρακολουθούσα τι γινόταν ε, σε σχέση με την εκστρατεία, σε σχέση με τα κοινωνικά μέσα και μέσω ενημέρωσης ε, και έπαιρνα την πληροφόρηση αυτή μέσω του διαδικτύου γρήγορότερα. Ξέρω ότι υπάρχει δυσκολία να πουλήσει κανείς έναν εκδότη σε μέσα σε θέματα ευρωπαϊκού χαρακτήρα, αλλά με αυτό του είδους ε, τα κοινωνικά μέσα θα μπορεί κανείς να προσφέρει περισσότερο τέτοια στοιχεία και να μπορέσει κανεί σε σχέση με το πρόγραμμα τηλεόρασης, τηλεοπτικό πρόγραμμα ή ραδιοφωνικό να υπάρχει μια ένταξη αυτών των ε, θεμάτων και να είμαστε πιο δραστήριοι μέσα στα πλαίσια των μέσων για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το κενό και να καταφέρουμε να προσανατηνώ σε σχέση με τα όσα τεκταίνονται. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και για αυτή την παρέμβαση. Ε, προτού σας εγκαταλείψω δυστυχώς, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Κοχμερίν, ε, γιατί θέλει να κάνει μια παρέμβαση σε σχέση με ε, την εισήγηση της κυρίας Καμπίνη. Νομίζω ότι θα είναι εμπλουτιστικό για τη συζήτησή μας. Έχετε το λόγο, κυρία Κόχμερη. Ε, ευχαριστώ. Μια ερώτηση θα ήθελα να διατυπώσω στην Λετήσια. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Μου άρεσε πολύ το ότι είσαστε. Είχατε εμβαθύνει στην ανάλυση τι είναι τα νέα μέσα ποια είναι η δημοκρατική συμμετοχή και τι είναι αυτή. Και θα ήθελα να ακούσω τον ορισμό σας των ευρωπαϊκών ειδήσεων. Τι είναι για σας ευρωπαϊκού χαρακτήρα ειδήσει. Είναι ειδήσει που, που δημιουργούν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι οι πληροφορίες που είναι ενδιαφέρουσες και αφορούν το σύνολο της Ευρώπης. Ποια, ποιος είναι ο ορισμός σας των ευρωπαϊκών ειδήσεων, ευρωπαϊκού χαρακτήρα ειδήσεων. Και έχω και μια ερώτηση προς εσάς λέει, συγγνώμη δεν μπορώ να διαβάσω εδώ το όνομα, αλλά εσείς είχατε πει ότι αναφέρατε ότι πληρώνοντα να πληρώνει κανείς για τις πληροφορίες, είναι κάτι που είναι ακόμα σημαντικό ω θέμα αρχής και ότι πρέπει κανεί να το δεχθεί για τον γραπτό τύπο και την ενημέρωση. Προβληματιζόμενοι τώρα σε σχέση με ένα περίεργο φαινόμενο, ίσως περίεργο φαινόμενο, το Σάββατο το βράδυ πριν από τις ε, εκλογές που είχαμε στη Γερμανία μια τηλεοπτική εκπομπή που δεν ασχολείται με πολιτικά θέματα καθόλου συνήθως σε μια πολιτικού χαρακτήρα συζήτηση υπήρχε ο Υπουργός Οικονομικών που και ηγέτες από όλα τα πολιτικά κόμματα επίσης και οι, όσοι ε, ε, συμμετείχαν έπρεπε να πληρώνουν για να συμμετέχουν στην, ε, στο opinion post, στην έκφραση απόψεων. Έπρεπε να καλέσουν ένα αριθμό ή να στείλουν ένα email και έπρεπε να πληρώσουν ένα τέλος στην, στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό. Μυριάδες συμμετείχαν που, που παρακολουθούσαν την εκπομπή και ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν για να εκφράσουν την άποψή τους ή να ψηφίσουν. Είναι ένα περίεργο, ασυνήθιστο φαινόμενο. Διερωτώμουν λοιπόν, τι είναι αυτό, τι μας λέει αυτό εμάς για το είδος του πώς παρουσιάζονται ειδήσει, για παράδειγμα σε σχέση με την πολιτική ζωή. Τι είναι αυτό. Είναι μια νέα, νέου είδους επιχείρηση αυτή, όπου πρέπει κάποιος να πληρώνει και οι ψηφοφόροι θα προσέρχονται σε αυξημένους αριθμούς για να συμμετέχουν. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σιλόγκα. Θα πρέπει να προεδρεύσει τώρα στην συνεδρίαση αυτή. Σας ευχαριστώ για την συμμετοχή σας. Okay. Well, uh, Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στον Σλανκό για να απαντήσω στην ερώτησή σας. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποια θα είναι η νέα μορφή των νέων μέσων και κανένας δεν ξέρει φαντάζομαι. Ναι, πραγματικά πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που προτίθενται να πληρώσουν για ε, ειδήσει υψηλού επιπέ... υψηλής ποιότητας. Και όπω σα είπα, μεταξύ 2000-2007 εργαζόμενοι εδώ σε μια οργάνωση που κάλυπτε τα θεσμικά όργανα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ήταν πολλοί που πλήρωναν για να έχουν τις πληροφορίες αυτές από βιομηχανικές ε, οργανώσεις, από ε, διοικήσεις κρατικές κλπ. Πλήρωναν και πολλά χρήματα μάλιστα για να ξέρουν τι γίνεται στην Ευρώπη. Και απαντώντα σε αυτά που είπε ο κύριος ε, και καταλαβαίνω, σημειώνω αυτό που είπατε για το θέμα ότι είναι πιο εύκολο τώρα, δηλαδή που οι Ιρλανδοί είπαν ναι, πολλά πράγματα διευκολύνονται. Ευχαριστώ. Κυρία Καμίνη, σας είχε αποτεθεί μια ερώτηση. Ναι, ο δικός μου ορισμός για τι είναι Ευρωπαϊκή Δύση. Τέσσερα πράγματα θα σας πω. Καταρχήν θα ήθελα να υπάρχουν ευρωπαϊκές συντακτικές ομάδες που προετοιμάζουν τις ειδήσεις αυτές όπου υπάρχει ο διάλογος μεταξύ των διαφορετικών προσεγγίσεων προς τις ειδήσει. Για τη συνεργασία με Ευρωπαίους δημοσιογράφους από παντού από όλη την Ευρώπη, μπορώ να σας πω ότι ο τρόπος της δημοσιογραφίας, η μέθοδος της δημοσιογραφίας στην Ιταλία, στην ε, Γερμανία, στη Γαλλία κλπ. διαφέρουν πάρα πολύ. Δεύτερον, να θεωρείτε ότι Ευρώπη σαν τη χώρα σας. Ίσως αυτή η πρόταση σας φαίνεται αντιφατική. Ελπίζω κανείς να με διορθώσει, αλλά θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη θεωρείται εξωτερική υπόθεση. Όχι, δεν είναι εξωτερική υπόθεση. Είναι η δική μας χώρα, το δικό μας συμφέροντα. Καλά και στι εξωτερικέ υποθέσεις έχουμε δικά μας συμφέροντα, αλλά πάντων. Αλλά δεν θα πρέπει να θεωρηθεί εξωτερική είδηση το τι ε, διαδραματίζεται στην Ευρώπη. Επίσης, θα πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο στο τοπικό επίπεδο, να μην έχουμε πάντα κατά νου τι Βρυξέλλες και ότι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ ή και στο Στρασβούργο που και που με χαρά μου άκουσα ότι πολλά από τα βραβεία που δόθηκαν δεν ασχολούνται με το τι γίνει διαγραμματίζεται στις Βρυξέλλες, αλλά σε τοπικό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι μπορούμε πραγματικά να καταστήσουμε την Ευρώπη λιγότερο εξωτερική είδηση, αλλά και πολύ περισσότερο σημαντική για την καθημερινή ζωή. Και μετά έχοντας υπόψη και την Ιρλανδική Προεδρία, ε, υπόθεση, συγγνώμη, την Ιρλανδική υπόθεση, θα πρέπει να θεωρήσουμε την Ευρώπη σαν μια ευκαιρία. Δεν είναι προπαγάνδα αυτό. Είναι ότι βλέπουμε τα καλά και δεν κατηγορούμε απλώς. Είναι εύκολο να κατηγορήσει κανένας. Αλλά αν μπορεί να δείξει κανένας ότι η Ευρώπη μπορεί να είναι χρήσιμη, θα μπορέσουμε να την επικρίνουμε κιόλας πιο καλά. Γιατί τη στιγμή η επικρίση κατά της Ευρώπης είναι πολύ χαμηλού επίπεδου και πολύ επιφανειακές και το είδαμε αυτό στα διάφορα δημοψηφίσματα που είχαμε για ε, την θεσμ... συνταγματική συνθήκη στη Γαλλία, στην ε, Ολλανδία και δύο φορές στην Ελλανδία. Και ήθελα να κάνω και μια παρατήρηση όσον αφορά το κατά πόσον οι ειδήσει αυτές ε, πρέπει να είναι ελεύθερες ε, ή να πληρώνει κανένας. Είναι επικίνδυνο να θεωρεί κανένας ότι η ειδήσει είναι χρησιμής μόνο για τις επιχειρήσεις. Οι ειδήσει είναι δημόσιο αγαθό και γι' αυτό θα πρέπει να είναι ελεύθερες και χωρίς πληρωμή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ίσως κάποιες ερωτήσεις και απαντήσεις να έχουμε για αυτό το θέμα πρώτα, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τον Ευρωπαϊκό χαρακτήρα δημοσιογραφ... για την δραστηριότητα ευρωπαϊκού χαρακτήρα δημοσιογραφία. Διαρωτώ αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό και να το συζητήσουμε έτσι. Και είναι ερώτηση προ εμά επίση. Μπορεί κανείς να κάνει λόγο για ευρωπαϊκή δημοσιογραφία αυτή αυτοτελώς. Δεν πρέπει να ορίσουμε τη δημοσιογραφία ως δημοσιογραφία πρώτα και μετά να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό κοινό χώρο αυτό είναι περισσότερο το ερώτημα που πρέπει να δημιουργηθεί αυτό ο Ευρωπαϊκό Δημόσιο Χώρο πρώτα. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Διότι δεν με ενδιαφέρει, δεν, δεν μου αρέσει αυτό ο όρο Ευρωπαϊκή Δημοσιογραφία. Προσπαθούμε επί χρόνια τώρα και το ασχολούμαστε με αυτό. Δεν νομίζω ότι θα λειτουργήσει σωστά έτσι. Κάποιε απόψει θα θέλω να ακούσω γι' αυτό πρώτα. Εσεί εσείς, εκεί παρακαλώ. Αυτό που λείπει ίσω είναι μια, ένας μεγάλος εκδοτικός οίκος διάδοσης αυτών των ευρωπαϊκού χαρακτήρα δημοσιογραφικών στοιχείων. Λέμε, διαβάσατε το άρθρο στη Γερμανία, στο Σπίγκερ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κανείς δεν ξέρει τις ίδιες εφημερίδες ή τα ίδια περιοδικά. Αυτό λείπει ένα κοινό έντυπο, ένα, μια κοινή εφημερίδα ή περιοδικό για τέτοιου είδους ειδήσει στο νέο τύπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άλλες απόψεις παρακαλώ. Εσείς παρακαλώ. Ένα από τα παραδείγματα που είναι αναγκαίο εδώ το ευρωπαϊκού χαρακτήρα ε, μέσο είναι το ότι έχουμε εδώ για παράδειγμα νικητές. Οποιοςδήποτε δεν βρίσκεται μέσα σε αυτό δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι έτοιμο για αυτό, αλλά χρειαζόμαστε αυτή την έκφραση για να διαφοροποιηθεί από την εθνική δημοσιογραφία η ευρωπαϊκή δημοσιογραφία. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, στο νέο, στα νέα έντυπα, δεν υπάρχει χώρος εδώ. Οποιοςδήποτε θέλει να ασχοληθεί με blogs ή Twitter και να κάνει σχόλια δεν μπορεί. Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω σε κάποιον σε, στην αίθουσα λέγοντα αν αυτή είναι καλή ερώτηση ή όχι. Θα έπρεπε να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση ή όχι και να γίνει η συζήτηση πολύ πιο ζωντανή και αξιόλογη με αυτόν τον τρόπο. Και νέοι bloggers, νέοι, νεαρής ηλικίας χρησιμοποιούν αυτού του είδους τις τεχνολογίες και μέσα για να είναι πολύ πιο αναζωογονημένες και ζωντανές οι συζητήσεις και πολύ πιο καρποφόρες σε σχέση με άλλα μέσα. Καλή παρατήρηση. Κύριε Σλάνκο, παρακαλώ, ανησυχώ πολύ να είμαι εγώ η φωνή των υπερσυντηρητικών, αλλά παρόλα αυτά, απαντώντας την παρατήρηση για τις δυσκολίες που υπάρχουν για την ευρωπαϊκή δημοσιογραφία το προφανέστερο είναι ότι δεν υπάρχει και η κοινή γλώσσα και το ξεχνάμε αυτό. Μιλάμε αγγλικά οι περισσότεροι και αυτό δεν είναι νομίζω εκείνο που μπορεί να υποκαταστήσει μια σωστή δημοσιογραφική γλώσσα έκφρασης. Και το άλλο θέμα είναι το περιεχόμενο των ευρωπαϊκών πολιτικών ε, τεκτενομένων που βρίσκεται στο επίπεδο των κρατών μελών ακόμα και όχι στο ευρωπαϊκό επίπεδο και τα θέματα τα κύρια σημασία όπω φορολογία ή εθνική άμυνα που παραμένουν στο επίπεδο κρατών μελών ω αρμοδιώτε, κυριαρχικά δικαιώματα δηλαδή. Και η προσοχή σχεδόν, ας το πω έτσι, σε αποκλειστικό, κατά αποκλειστικότητα είναι στις ε, εθνικές πρωτεύουσες, στα κράτη-μέλη για τέτοιου είδους ειδήσει και τι γίνεται με τις ευρωπαϊκού χαρακτήρα ειδήσει. Δεν είμαι βέβαιος ότι πρέπει να αλλάξει αυτό, γιατί η βάση, ε, τα θεμέλια των δημοκρατικών πολιτικών είναι τα κράτη, τα κράτη-μέλη και δεν έχουμε ευρωπαϊκό κράτος ως σύνολό του αυτή τη στιγμή. Και έτσι σε σχέση με την ε, κοινότητα που βλέπουμε και τον τύπο, σε εθνικό επίπεδο μπορεί να κινηθεί περισσότερο. Δεν μπορώ να δω με ποιον άλλο τρόπο θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα υποκατάστατο. Ευχαριστώ δύο λόγια μόνο για την παρατήρηση καλού, καλής και κακής δημοσιογραφίας. Συμφωνώ, είναι πολύ πιο εύκολο να έχουμε καλή δημοσιογραφία αν τηρεί κανείς τους παραδοσιακούς κανόνες της δημοσιογραφίας. Και αν δεν αφήσει κανείς σε ένα ανοιχτό πλαίσιο τα πάντα να είναι ελεύθερα και χωρίς έλεγχο. Και για τις συνεισφορές ε, και που είναι εύκολο να γράψει κανείς ε, ιστορίες ε, για ειδήσει που δεν χρειάζεται μεγάλη ε, δουλειά για τεκμηρίωση και σε σχέση με ε, το έπαθλο πραγματικά που με εντυπωσίασε σε σχέση με ε, γενικούς όρους η δουλειά αυτή. Αν όμως δει κανεί όχι μόνο θέματα που ο ίδιος αλλά και άλλοι είχαν να συντάξουν και έπρεπε πολύ μεγάλη δουλειά για τεκμηρίωση να γίνει και πολλά χρήματα να επενδυθούν από πλευρά των εκδοτών Πώς θα μπορούσε κανείς ε, να το κάνει αυτό με τους νέους κανόνες για τα νέα μέσα τύπου, όπου δεν, υπάρχει εδώ, ε, δεν υπάρχουν έσοδα όσον αφορά για παράδειγμα <coughs> διαφημίσεις. Δυστυχώς τα χρήματα διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο όταν κάνουμε λόγο για την ποιότητα της δημοσιογραφίας. Και επίσης για να διασφαλίσουμε την αναγκαία ανεξαρτησία και την αναγκαία, ας το πω έτσι, εξέταση των στοιχείων, το χτένισμά τους, ε, για να μπορέσουμε να είμαστε σε υψηλή ποιότητα δημοσιογράφοι. Και σε αυτό το οποίο αναφέρθηκε από τον Γερμανό που παρενέβη για το ευρωπαϊκό δημόσιο χώρο, σίγουρα η γλώσσα είναι μείζον πρόβλημα που δεν έχουμε μια κοινή γλώσσα. Αν δει κανείς όμως το τι γίνεται το ότι έχουμε μία γλώσσα που μιλάνε όλοι τα αγγλικά και που παραμορφώνεται και αν γίνεται κάποια ζημιά και από γλωσσικής πλευράς πλέον. <clears throat> Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έγιναν προσπάθειες πρόσφατα να συνταχθεί, να καταρτιστούν τα ευρωπαϊκά, ευρωπαϊκού χαρακτήρα ε, έντυπα. Πριν από 15 χρόνια ένα έντυπο The European που εξαφανίστηκε. Δεν υπήρχε αρκετό ενδιαφέρον από πλευράς ε, των πολιτών για ένα τέτοιο έντυπο. Έχουμε εδώ ένα ε, εβδομαδιαίο έντυπο, η Ευρωπαϊκή Φωνή, the European Voice, αλλά στοχοθετημένα ε, δημοσιεύει για ανθρώπους που δουλεύουν στις Βρυξέλλες. Και απλά και μόνο θα ήθελα μία παρατήρηση να κάνω από πλευράς κάποιου που επί χρόνια συμμετέχει σε αυτά τα πλαίσια παρατήρησα ότι ενώ οι διαδικασίες ολοκλήρωσης συνεχίστηκαν και προόδευσαν και θα αρχίσει να ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας και αυτό θα διευρύνει την πρόοδο σίγουρα, υπάρχει μια ένας διαχωρισμός ακόμα ισχυρότερος και εντονότερος όσον αφορά τις ευρωπαϊκές ειδήσει ε, πώς διαχέονται και πώς ε, καταλήγουν στο, στο, στο εθνικό κοινό, στα κράτη-μέλη. Όταν ξεκίνησα εδώ και πιθανότατα επειδή το θεσμικό πλαίσιο ήταν πιο εύκολο. Γράφαμε για οικονομικά κυριότερα θέματα όπως την ΚΑΠ, την κοινή αγροτική πολιτική, την χαλιβουργία, τα αυτοκίνητα, την αυτοκινητοβιομηχανία κτλ. Ήταν κάτι που συσχετιζόταν ουσιαστικά στα ίδια προβλήματα. Τώρα βρίσκω ότι με την τελευταία διεύρυνση αλλά και ήδη ξεκινώντας πριν από αυτήν η όσοι δουλεύουν στις Βρυξέλλες ως δημοσιογράφοι παίρνουν πολύ περισσότερο μια εθνική προσέγγιση, μια εθνική θέση ε, τοποθέτηση. Δεν είναι αυτό αναγκαστικά μια αντίφαση λόγω του επίπεδου ολοκλήρωσης που έχουμε ήδη επιτύχει στην Ένωση. Και αυτό είναι αρκετά φυσικό θα έλεγα, να υπάρχουν περισσότερες τριβές που αποκαλύπτονται και εθνικά συμφέροντα να αντικρούονται και να βρίσκονται αυτά στο προσκήνιο πλέον και να αποκαλύπτονται νομίζω είναι μια φυσική εξέλιξη των πραγμάτων αυτή. Και είναι κάτι το οποίο θα καταστήσει περισσότερο δυσχερές δύσκολο να καταλήξουμε στην έννοια της ε, ευρωπαϊκού χαρακτήρα κοινή ε, ας το πω έτσι, αρένας. Σας ευχαριστώ. Θα έρθω σε εσάς, θα λάβετε τον λόγο. Αλλά η κυρία Κοχμερή νομίζω θέλατε να παρέμβετε παρακαλώ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο. Δυστυχώς έχω ανηλυμένες υποχρεώσεις και θα πρέπει σε λίγα λεπτά να φύγω, αλλά παρόλα αυτά μια παρατήρηση ακόμα θα ήθελα να κάνω, διότι μια ερώτηση διατυπώθηκε για τη δημοκρατική συμμετοχή. Θα ήθελα, μου αρέσει η ιδέα και ο ιδεαλισμός ε, και τα ιδανικά από πλευράς ε, της ομίγυρης για τις νέες δυνατότητες των νέων μέσων. Θα ήθελα να διατυπώσω το ερώτημα. Αυτό δεν είναι, ας το πω έτσι, ένας καταμερισμός, μια, ένας διχασμός της κοινωνίας σε μια ελίτ όσον αφορά την ενημέρωση που ενδιαφέρεται για συγκεκριμένου είδους πληροφορίες από πλευράς περιεχομένου για συμμετοχή στη συζήτηση, ένα πολύ χαμηλό ποσοστό αν δει κανεί τα θέματα δημοκρατίας και το δικαίωμα να ψηφίζουν και να συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες όλοι, τουλάχιστον όλοι πάνω από τα 18 έτη. Δεν υπάρχει μεγάλο χάσμα, μεγάλο χάσμα δημοκρατικότητας θα έλεγα. Δεν καλύπτεται εδώ αυτό από τα νέα μέσα. Αλλά η δημοκρατική συμμετοχή δεν θα πρέπει να, συμμετα... να αυξάνεται ε, με τη συμμετοχή σε αυτά τα πλαίσια. Είναι ίσως μια ιδεαλιστική αφελής προσέγγιση αυτή. Τι συμβαίνει. Απλώς διατυπώνω το ερώτημα για να το απαντήσετε αν γίνεται. Και αυτό το οποίο αναφέρθηκε για το BBC ότι 75% των νεαρών ανθρώπων δεν μπορούν να φανταστούν να ζουν χωρίς το διαδίκτυο, χωρίς το ίντερνετ. Εγώ είμαι πολύ πάνω από αυτό το όριο, αλλά παρόλα αυτά και αυτό είναι σημαντικό για τη ζωή μου. Όμως ποιο είναι το ίντερνετ και το να είναι αυτό το πιο σημαντικό στη ζωή κάποιου. Δηλαδή τι, για τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μήπω υπάρχει εδώ ένα χαμηλό ποσοστό όσον αφορά την, ε, το περιεχόμενο αυτό. Τι είναι εκείνο που καθιστά α, ε, χωρίς δυνατότητα υποκατάσταση στο ίντερνετ αναντικατάστατο στη ζωή των ανθρώπων. Τι γίνεται σε σχέση με τη δημοκρατική συμμετοχή. Το ίδιο το μέσο δεν είναι η απάντηση στο ερώτημα. Πρέπει να ξαναπροβληματιστούμε ίσως για τον τρόπο τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τη σημασία, τη σπουδαιότητα της δημοκρατίας και με αυτό να δημιουργήσουμε μεγαλύτερα πλαίσια, ευρύτερα πλαίσια συμμετοχής ε, δημοκρατικά. Ευχαριστώ. τώρα εκεί, εσείς παρακαλώ, εκεί πίσω όνομά μου Μάριος Γκαρέλα. Είμαι νέος δημοσιογράφος, αλλά και ακολουθώ και ε, εργασία λομπιίστα μέσω της δραστηριότητά μου. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το οποίο αναφέρατε. Ευρωπαϊκού χαρακτήρα δημοσιογραφία ή ευρωπαϊκός κοινό χώρος. Βλέπω μια καλά οργανωμένη για παράδειγμα εθνική εφημερίδα, γερμανική, ιταλική, γαλλική και σε σχέση με του δημοσιογράφου τη Βρυξέλλε που ανταποκρίνονται όσον αφορά το μεγαλύτερο μέρο τη δημοσιογραφική δουλειά ε, για την εφημερίδα ή το μέσο που βρίσκεται στην εθνική πρωτεύουσα. Δημοσιογράφοι ανταποκριτέ, θα σα πούν δεν υπάρχει αρκετό χώρο για θέματα ευρωπαϊκά. Οι εκδότε του δεν ενδιαφέρονται για τα ευρωπαϊκά θέματα. Και αυτοί οι εκδότε είναι τα άτομα που βρίσκονται για παράδειγμα σε σχέση με την ηλικία. Όσοι έρχονται ε, συμμετέχουν στην ε, σε αυτές τις διαδικασίες, δεν έχουν όμως ε, πρόσβαση στα όσα γίνεται, γίνονται στις Βρυξέλλες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό είναι κάτι που διευρύνεται όλο και περισσότερο σε σχέση με τους εκλογείς. Κάθε πέντε χρόνια τους ζητάνε να συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές και δεν γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται και τι, τι είναι αυτά τα ευρωπαϊκά θέματα. Για μένα αυτό θα αλλάξει όταν οι ανταποκριτές στις Βρυξέλλες θα έχουν μεγαλύτερες ευκαιρίες ε, και όταν θα υπάρχουν περισσότεροι δημοσιογράφοι ανταποκριτές για την ίδια αλυσίδα ή τηλεοπτικό σταθμό ή μέσο, ε, τότε μπορεί να συνεργαζόμενοι αυτοί να δημιουργήσουν ένα ευρωπαϊκό κοινό χώρο διότι δεν θα χρειάζεται να ταξιδεύουν ε, σε σχέση με τις χώρες. Θα μπορούν να, γνωρίζουν μέσω των ειδήσεων τι γίνεται και να έχουν αρκετή πληροφόρηση, ικανή πληροφόρηση για να μπορούν να ψηφίζουν στο τέλος. Αυτό είναι ο ευρωπαϊκού χαρακτήρα ε, δημοσιογραφικός χώρος. Να γνωρίζουν τι γίνεται στην Ευρώπη, να είναι ενημερωμένοι και εξοικειωμένοι με αυτά. Σας ευχαριστώ. Εσείς εδώ μπρος. Uh, just a couple a couple of questions for, for Mr. Μερικές ερωτήσεις για τον κύριο Η μία είναι η τίνος πρόκειται το, για το θέμα το διασυνοριακό, Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο κλπ. Μετά το θέμα της κρατικής χρηματοδότησης για την δημοσιογραφία η Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώ ε, χρηματοδοτεί το Euronews. Θα συμφωνούσατε να προσθέσει και χρηματοδότηση για τα νέα μέσα ενημέρωσης, για, τα, για το διαδίκτυο κλπ. για να δημιουργηθεί το νέο αυτοκοινό Ευχαριστώ, θα επανέλθω, λέει ο Πρόεδρος. Παρακαλώ, μία ακόμα ερώτηση. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, εντάξει. Οκταβιά Ζωρά από τη Ρουμανία. Είμαι δημοσιογράφος και είμαι και επικουρικός ε, καθηγητής οικονομικών στην, ε, στο Βουκουρέστι. Θα ήθελα να κάνω δύο-τρία σχόλια για δύο-τρία θέματα που μου έκαναν εντύπωση όταν τα έκοσα εδώ. Ένα από τα ερωτήματα που μου έκανε εντύπωση ως οικονομολόγος είναι το γεγονός ότι το προϊόν της δημογραφίας θα πρέπει να θεωρηθεί κοινό αγαθό δημόσιο αγαθό και αυτό θα πρέπει να μην κοστίζει τίποτα. Μεταξύ επαγγελματιών, κάθε φορά που είμαι σε επαφή με τέτοιες ομάδες, τα προϊόντα τους είναι όλα υπέρ, ε, ε, είναι το, το, επίκεντρο της ζωής ή, όταν είμαι μεταξύ γιατρών, τα ε, ιατρική η ιατρική επιστήμη είναι γενικό αγαθό, όταν μεταξύ τραπεζιτών τα χρήματα, όταν είμαι μεταξύ δημοσιογράφων, το ίδιο για τις ειδήσει. Εγώ δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να είναι όλα αυτά α, ελεύθερα, γιατί σχολιάζοντας την ε, παρουσία της κυρίας Γκαμπίνη, έχω μία συμβουλή για εκείνους που θεωρούν ότι η δημοσιογραφία είναι ένα κοινό αγαθό. Εγώ έχω να σας πω, αν θέλετε τα αγαθά σας να είναι δωρεάν, δώστε μου του δωρεάν. Μην μου ζητείτε να πληρώνω ούτε φόρους, ούτε να σας επιδοτώ άμεσα. Δεν χρειάζομαι να πληρώνω φόρος, να σας πω. Θα ήμουν ευτυχής και χωρίς. Μετά, κάτι που έθιξε ο κ. Λέκεγκάρτ. Είπατε ότι είσαστε φιλελεύθερος με θέμα, ιδίως όσον αφορά τα ε, θέματα των ΜΜΕ. Έχω την εντύπωση ότι προσπαθώντας να επιληθεί το πρόβλημα της παρέμβασης μεταξύ των εκδοτών ή των ιδιοκτητών των ε, μέσων ε, μαζικής ενημέρωσης και της παρέμβασης, αν παρέμβει μια κυβέρνηση, τι θα λυθεί. Δεν θα ήθελα να υπάρχει ένα μέσο του οποίου η κυβέρνηση υπαγορεύει το τι θα πρέπει να γίνει, τι δεν θα πρέπει να κάνει και να πει. Νομίζω ότι η αγορά για τους δημοσιογράφους είναι εκείνη που θα ε, κυρώνει κακή συμπεριφορά. Γιατί οι δημοσιογράφοι μπορούν να πάνε από τον έναν εκδότη στον άλλον εκδότη να έχουν δικέ του ε, απόψει. Δεν χρειάζεται νομίζω παρέμβαση κυβέρνηση, γιατί μια παρέμβαση κυβερνητική σημαίνει ότι ε, προσπαθεί έτσι να φιλτράρει, αν θέλετε, τα μηνύματα που περνάνε. Τρίτο σχόλιο. γιατί ότι θα πρέπει κανένας να ασχολείται με εθνικά θέματα για να μπορέσει να πάρει ένα βραβείο εδώ. Εγώ προσωπικά έγραψα ευρωσκεπτισχιστικά για το δημοψήφισμα ε, για την Ιρλανδία και πήρα το βραβείο στη Ρουμανία. Σε ευχαριστούμε. Κάποιοι παραπάνω ακόμα να παρέμουν και μετά θα περάσουμε στο πάνελ. Εσείς εκεί και μετά εσείς από παραδίπλα. Μ' ακούτε, μπορώ να παρέμβω. Εντάξει. Από τη Σουηδία ε, προσέρχομαι. Από ραδιοφωνικό σταθμό. Δεν ήθελα να σχολιάσω αυτό το οποίο ανέφερε η κυρία Γκαμπίνη για του ευρωπαϊκού χαρακτήρα δημοσιογραφία και μίντια. Είναι ενδιαφέρον εγχείρημα αυτό που έχει ξεκινήσει για τα ευρωπαϊκά μέσα, αλλά ακούγεται και ελιτιστικό ίσως ταυτόχρονα, αλλά και ευρωσκεπτικιστές ε, θα μπορούσαν πολύ εύκολα να συμπεριληφθούν. Δεν νομίζω ότι πρέπει να έχει κανείς μια αρχικά θετική θέση. Δεν χρειάζεται αυτό για να ενδιαφέρεται για ευρωπαϊκά θέματα. Τα θέματα συμμετοχής είναι σημαντικά. Ευχαριστώ εσείς. Παρακαλώ. Από πλευράς ε, Ιρλανδίας ε, από την οποία έρχομαι. Χαίρομαι και σέβομαι την ε, άποψη για την ε, ελεύθερη δημοσιογραφία και για την δημόσια χρηματοδότηση. Υποθέτω ότι θα υπάρχει η χρηματοδότηση αυτού του είδους δραστηριοτήτων και είναι κάτι που θα είμαι πολύ σύντομο στην παρέμβασή μου. Αφορά το διαδίκτυο και καθώς προέρχομαι ε, το θέμα της δημοσιογραφίας είναι ότι εξ ορισμού το ίντερνετ δεν διαχωρίζει και δεν διαφοροποιεί τα πράγματα ούτε έχει διαχωριστικές γραμμές είναι ας το πω έτσι χωρίς επιλογή ή χωρίς ε, κάποιες προδιαγραφές ένα πλαίσιο έκφρασης το θέμα είναι ότι για παράδειγμα όταν υπήρχε, υπήρχαν ψήθυροι ότι είχε αποβιώσει ηθοποιός ε, του Hollywood και όλα αυτά καταδείχθηκαν στη συνέχεια ότι ε, δεν ήταν ακριβώς όπως είχαν αρχικά αναφερθεί. Είναι σημαντικό εδώ να δει κανείς ε, την δημοσιογραφία που πρέπει να εξετάζει τα πράγματα πρωτού διαχέει ειδήσει και να χτενίζει το περιεχόμενο. Τώρα εδώ σε σχέση με την δυνατότητα να εκφράζονται περισσότερη άποψη, αυτό είναι δεδομένο. Όμως ούτε και από αυτό το πλαίσιο αναβαθμίζονται κάποιες απόψεις ε, και μέσω των διαφορετικών blog ε, δεν υπάρχει, ας το πω έτσι, εμπλοκή σε σχέση με κάποια θέματα. Απλά και μόνο επίπεδο συζήτησης είναι στο επίπεδο των blogs. Πολλά πράγματα τα οποία για παράδειγμα όσον αφορά την πληρωμή τελών πνευματικών ε, δικαιωμάτων ε, ή ε, Μέχρι ποιο, ποιο βαθμό νομίζετε ότι θα μπορέσει αυτό να προχωρήσει μέχρι ότου υπάρξουν προδιαγραφές και ρυθμιστούν αυτά τα πλαίσια ή είναι δυνατόν εδώ να υπάρχει ένα χαλαρότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα δραστηριοποιούνται όσοι εμπλέκονται χωρίς να πληρώνουν. Ευχαριστώ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις Νομίζω δεν ξέχασα κανέναν τελευταίο εσείς εκεί παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω στον κύριο Σταβένο, συγγνώμη για την προφορά του ονόματός σας, είμαι Ισπανίδα, δεν είμαστε ιδιαίτερα ε, προσοντούχοι στις γλώσσες. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που θα ήθελα να ε, θίξω. Θα ήθελα μια παρατήρηση να κάνω. Φοβούμαι ότι πραγματικά διαφωνώ πρέπει να πω με αυτό το οποίο είπατε, ότι τα νέα μέσα κοστίζουν χρήματα και πρέπει να επενδυθούν κονδύλια για να επιβιώσουν αυτά τα νέα μέσα. Εγώ βρίσκομαι εδώ λόγω του ότι συμμετείχα μέσω blog και αυτά δεν κοστίζουν καθόλου, είναι δωρεάν και παίρνω και βίντεο μέσω, της, ε, ε, μέσω παρόχου που ελεύθερα δωρεάν παρέχει αυτό το υλικό. Επίσης και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μηδενικές, ε, μηδενικά τέλη, δωρεάν πάλι και έχω και κάρτες ταχυδρομικές που κατασκευάζω εγώ ίδια και διαχέω, πάλι μηδενικές δαπάνες εκεί, δωρεάν. Αλλά η ερώτηση προς την κυρία Γκαμπίνη και η παρατήρηση είναι επειδή το πώς θα είναι δυνατόν το θέμα των χρημάτων εδώ να διαφοροποιηθεί. Είμαστε δημοσιογράφοι, δεν μπορούμε δωρεάν να ζούμε χωρίς μισθό. Πρέπει να πληρώνουμε και τους λογαριασμούς, λογαριασμούς μας. Και αυτό είναι το πρόβλημα που έχω με τον blog μου. Δεν μπορώ να ζω από αυτό, δεν μπορώ να εισπράξω χρήματα από τη δραστηριότητα, μου ως μπλογγίστας. Πρέπει να, να έχω μια άλλη δραστηριότητα για να καλύπτω τα, τις δαπάνες μου. Ίσως θα πρέπει να το δούμε αυτό και είναι μια πρόταση Νομίζω καλή πρόταση θα ήταν να μπορούμε να εισπράττουμε χρήματα από ε, ειδήσει αναβαθμισμένης ποιότητας, υψηλής ποιότητας. Χρειαζόμαστε όμως ε, τις ειδήσει αυτές ε, και το γνωρίζω ότι στην Ισπανία υπάρχει έλλειψη ειδήσεων από πλευράς του ευρωπαϊκού επίπεδου από την Ευρώπη οι κυριότερες εφημερίδες στην Ισπανία δεν ε, ε, έχουν πολλά για τα, ε, τις ευρωπαϊκές ειδήσει και καταλήγουν έτσι άνθρωποι στο blog και έτσι μέσω του blog επικοινωνούμε. Και εδώ τα νέα μέσα του τύπου δεν εισπράττουν χρήματα, δεν έχουν έσοδα και έτσι και οι πολίτες έχουν πρόβλημα. Πώς δηλαδή να συμμετάσχουν μέσα σε αυτά τα πλαίσια των νέων μέσων του τύπου όταν δεν υπάρχει ας το πω έτσι συνιστόσα της διασφάλισης των εσόδων. Καλό θα ήταν να μπορούσαμε χρησιμοποιούσαμε, να δημιουργούσαμε ένα δίκτυο εδώ και τώρα. Ε, οι εθνικοί ε, ε γιατί να μην μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο και να συνεργαστούμε μεταξύ μας. Εντάξει, σωστό, δεν έχουμε ακόμα μια κοινή γλώσσα, εντάξει δεν μπορούμε να εργαστούμε διότι εντάξει εγώ μιλάω διάφορες γλώσσες και είμαι σίγουρη ότι και άλλοι εδώ μιλάνε διάφορες άλλες γλώσσες πέρα από τα αγγλικά. Χρειαζόμαστε όμως, μια και είμαστε δημοσιογράφοι, να μιλάμε ξένες γλώσσες. Να δώσουμε συνέχεια λοιπόν σε αυτό. Ευχαριστώ για την πρότασή σας. Πρέπει να κλείσει η συνεδρία σε πέντε λεπτά. Θα πρέπει να περάσουμε στο πάνελ τώρα Υποσχέθηκα όμως τον κύριο εκεί κάτω, εσείς μπορείτε σε μισό λεπτό να κάνετε την παρατήρησή σας, παρακαλώ. Εσείς ε, κύριε εκεί πίσω. Εντάξει, σας ευχαριστώ λοιπόν. Τότε περνάμε στα, στους όσους συμμετείχαν στο πάνελ, θα έχουμε τις καταληκτικές παρατηρήσεις, ο κύριος Λάγκο. Ένα άλλο επιχείρημα να χρησιμοποιήσω για τις ειδήσει έναντι πληρωμής. Πιστεύω το γεγονός ότι οι εφημερίδες εισπράττουν για το, τις ειδήσει που παρέχουν δημιουργεί έναν υγιή δεσμό, ένα κρίκο μεταξύ των δημοσιογράφων και των αναγνωστών. Όταν παράγει κάποιος κάτι που κάποιος θα πληρώσει γι' αυτό ε, τότε δημιουργείται ένα υγιές περιβάλλον, να το πω έτσι, και υγιής σεβασμός για σας που παράγεται αυτήν την είδηση και σε σχέση και με τους αναγνώστες. Δεν είναι, ε, νομίζω, να εκπλήττει κανέναν ότι είναι πολύ χαμηλότερης ποιότητας τα δωρεάν έντυπα, ή δωρεάν εφημερίδες. Δεν είναι μόνο ότι έχουν λιγότερα χρήματα για να παράγουν αυτές οι ειδήσεις, αλλά αν δεν εισπράττεις για αυτό το οποίο παράγεις, ε, τότε το επίπεδο θα είναι διαφορετικό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για να απαντήσω κάποιες ερωτήσεις εγώ ίδιος. Νομίζω το θέμα πληρωμής ε, και το θέμα του funding, state funding, κρατικής, ε, ας το πω έτσι, επιχορήγησης ή πληρωμής. Νομίζω παράδοξο είναι μια αντίφαση που υπάρχει. Αν πραγματικά πιστεύετε στην ελεύθερη αγορά όπως εγώ και την ικανότητα της ελεύθερης αγοράς να επιλύει προβλήματα, τότε θα αντιληφθείτε ότι σε σχέση με τις ε, χώρες της Ευρώπης ε, υφίσταται πρόβλημα με τον ελεύθερο ε, την ελεύθερη δημοσιογραφία ανάλυσης και έρευνας Τώρα, σε σχέση με την πολιτική εμπλοκή, όχι μόνο σε σχέση με το έργο φυσικά της δημοσιογραφίας, αλλά για τη συλλογή εσόδων, μόνο για τη δανέζικη εμπειρία μπορώ να κάνω λόγο φυσικά και γνωρίζω ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς αυτή την πείρα πανευρωπαϊκά, όμως σε ευρωπαϊκό επίπεδο χρειαζόμαστε κάποιες λύσεις, χρειαζόμαστε έσοδα. Δεν γίνεται να επιληθούν τα προβλήματα χωρίς ε, έσοδα, χωρίς εισπράξεις, ε, όπως είπε και ο προλαλής σας. Δεν έχω το ιδανικό εργαλείο και μέσο να πω τι θα μπορούσε καλύτερα να λειτουργήσει, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτό το γεγονός για να την απαντήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις. Τώρα, ίσως ε, να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση τώρα και θα αφήσω τώρα τον, τον λόγο να τον λάβετε εσείς για να ολοκληρώσετε από πλευρά σας. Σύντομα, δεν ζητούμε να υπάρξει επιχορήγηση ή να υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης προϊόντων δωρεάν στην αγορά. Το αντίθετο, αν κάποιος είναι πρόθυμος να πληρώσει για ένα προϊόν, τότε υπάρχει η εγγύηση ότι καλής αξίας θα είναι αυτό το αντιθετο αν καποιος ειναι προθυμος να πληρωσει για ενα προιον τοτε υπαρχει η εγγυηση οτι καλή αξία θα ειναι αυτο το οποίο πληρώνεται και αγοράζεται. Τώρα, για την δημόσια τηλεόραση και του τηλεοπτικούς σταθμούς, εδώ είναι ένα διαφορετικό στοιχείο. Πληρώνονται από δημόσια έσοδα προς όφελος του κοινού, για το συμφέρον του κοινού, για να διατίθεται πληροφόρηση από ανεξάρτητους ε, δημόσιους δημοσιογράφους και ενημέρωση. Αυτό θα έπρεπε να είναι και πρέπει να είμαστε, αυτό πρέπει να συμβαίνει και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί να διασφαλίζουμε ότι αυτό θα γίνεται. Και είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με τον ρόλο των δημόσιων σταθμών σε αυτή τη συγκυρία και χρονική συγκυρία όπου υπάρχουν τόσες διαφορές και υπάρχει μεγάλη, μεγάλος ανταγωνισμός Μπορεί να είναι θετικό αυτό. Αν έχει κανείς ε, ένα καλώς ε, λειτουργούν ε, σύστημα δημοσίων υπηρεσιών, αυτό μπορεί να είναι υπέρ του κοινού, υπέρ των πολιτών. Και αυτό δεν αφορά μόνο τα θέματα για το όφελος ε, που αφορούν την ερώτησή σας, για τα έσοδα, αν που θα, τα κονδύλια που θα διαχέονται για να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε την κάλυψη ευρωπαϊκών ειδήσεων. Το Euronews είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Αν το δει κανεί έτσι, είναι θα έλεγα δύσκολο να διακριβώσει κανείς ε, την ε, ε, δημοσιογραφική, ας το πω τον δημοσιογραφικό πυρήνα της δουλειάς τους. Είναι κάτι το οποίο έχει εισαχθεί από κάποιους ε, για να υπάρξουν δημόσια κονδύλια που θα διασφαλίσουν για αυτή τη δραστηριότητα που ακολουθούν από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με αυτού του είδους τις δραστηριότητες. Και όσον αφορά την ε, EuroTV και κάνω λόγο και για τους, ε, την Ένωση των ε, Ευρωπαίων Ανταποκριτών στις Βρυξέλλες, πιστεύουμε ότι υπάρχει κίνδυνος εδώ. Αν θεσμικά όργανα ξεκινήσουν κάτι και εμπλακούν σε κάτι, το οποίο θεωρείται αρχικά ως ανεξάρτητη δημοσιογραφία, στο τέλος τέλος όμως χρηματοδοτείται από κάποιο θεσμικό όργανο και λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε κόμμα, κάθε κοινοβουλευτική ομάδα που εκπροσωπείται ανάλογα με το ποσοστό τους ε, που τους αναλογεί ε, επηρεάζουν. Αυτό δεν είναι ε, ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Είναι κάτι το επιζήμιο κιόλα για εκείνους τους δημοσιογράφους που προσπαθούν στο σωστό επίπεδο και ύψος των περιστάσεων να ασκήσουν το επάγγελμά τους. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ κύριε Καμπίνη. Ναι, για τα χρήματα. Ίσως το καλύτερο είναι να είναι κανείς δημιουργικός και να αρχίσει να συμπεριλαμβάνει στις σχολές δημοσιογραφίας και μαθήματα για τα πώς συλλέγει κανένας χρήματα. Για να είμαστε πιο σοβαροί, η παρατήρηση από τον Σουηδό συνάδελφο. Ίσως δεν με κατανοήσατε εγώ, θα ήθελα πιο κριτικές ε, ειδήσει για την Ευρώπη. Νομίζω ότι για την δημοκρατική υγεία της κοινωνίας είναι καλό να υπάρχουν κριτικές φωνές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί κανένας να καταδεικνύει ότι δεν είμαστε τέλειοι. Σίγουρα η Ευρώπη δεν είναι τέλεια. Και φαίνεται αυτό ξεκάθαρα όταν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έρχεται σε μια αίθουσα γεμάτη δημοσιογράφους και ζητά συγγνώμη ότι τα 27 κράτη-μέλη δεν μπορούν να συμφωνήσουν πάνω σε κάτι. Δεν είναι τέλεια λοιπόν η Ευρώπη, αλλά αυτό που θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε είναι πώς θα μπορούμε να είμαστε κριτικοί πιο ευφυώς να χρησιμοποιούμε τη δυνατότητα να ερχόμαστε εδώ, να συζητάμε με τους πολιτικούς, να μιλάμε με τις Βρυξέλλες, αν θέλετε, να κατανοούμε ποιοι είναι οι μηχανισμοί και ποια είναι τα προβλήματα που θα πρέπει να μεταβάσουμε στα ακροτήριά μας. Όπως είπε και η Ισπανίδα συνάλφος, αυτό είναι πρόβλημα για όλους, γιατί δεν είναι κανένας ικανοποιημένος. Δεν είναι μια κατάσταση στην οποία όλοι κερδίζουν, τουναντίον όλοι χάνουν. Δεν υπάρχουν χρήματα για μας, οι συντάκτες δεν μας δίνουν αρκετό χώρο, οι καταναλωτές, οι πολίτες δεν έχουν αρκετές ειδήσει. Ένας φαύλος κύπλος θα έλεγα. Εγώ θεωρώ ότι είναι ευκαιρία τα νέα μέσα, ε, καταλαβαίνετε συμφωνείτε όλοι μαζί μου, αλλά θα ήθελα να σας καλέσω όλους να προσπαθήσετε να πειραματιστείτε όπως το κατανοείτε είτε μέσα των νέων μέσων είτε των παλιών, δεν έχει σημασία. Θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερες ευρωπαϊκές ειδήσει πάντως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Καμπίνη. Πρέπει να κλείσουμε εδώ. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερο χρόνο εδώ και τώρα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα, πάρα πολύ σημαντική συζήτηση. Θα σας ευχαριστήσω που ήρθατε εδώ και συμμετείχατε σε αυτή τη συζήτηση και σας διαβεβαιώ ότι ήταν πάρα πολύ πιο καλά εστιασμένοι από πολλές, πολλές συζητήσεις του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Excuse me, just an organizational thing. We have um, a lunch at 12.30 organized for the national winners, to which you're welcome. And from 12.15 onwards, the reimbursement process will, will start and people will be guided to the CAS to receive their... Η στροφή των εξόδων θα αρχίσει τώρα. Οι συνάλληλοι θα ασχοληθούν με αυτό. 12 και 4 και λοιπά. Το γεύμα θα είναι στο εστιατόριο ε, του, των βουλευτών θα σας οδηγήσουν και εκεί που πρέπει να πάτε.